Okay. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Uh, it's time to start our meeting. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας σε τρία μέρη. Δηλαδή Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 πρωί και απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, η μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να δεχθούμε την μερίσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Δεν βλέπω κάποιος να θέλει να σχολιάσει την μερίσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Ουδεμία. άρα πάμε γρήγορα και εύκολα. Πάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Της 20 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2015. Αν δεν έχετε σχόλια, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Ωραία. μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας. Έκθεση που δεν θα μας παρουσιάσει αυτή τη φορά η κυρία Γκρίφιν, αλλά η κυρία Μούντι, μέσα σε ένα λεπτό, μάλλον θα τζώσω σε ένα λεπτό. Η έκθεση αυτή βασίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν του 2015 για μια νέα συμφωνία για τους ε, κατάλληλες ενέργειες. Βλέπετε ότι προχωρούμε προς την Ενεργειακή Ένωση βήμα-βήμα. Θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση συνδέεται στενά με την έκθεση του κ. Λάγκεν για το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού και τέλο πάντων γενικώ για το σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας και είναι μια έκθεση αυτή την οποία θα συζητήσουμε σε 45 λεπτά περίπου. Αυτές οι δύο εκθέσεις είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η δεύτερη φορά κυρίως στην αγορά ηλεκτρισμού, όχι τόσο το φυσικό αέριο. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο πίσω και να πάμε στην έκθεση της κυρίας Γκρίφιν γιατί δεν έχει αλλάξει. Στα ακτρέ είναι η κυρία Γκρίφιν, παρότι δεν είναι εδώ σήμερα. Η συνάδελφος κυρία Μούντι, παρακαλώ να λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Δυστυχώς ε, η Τερέσα Γκρίφιν δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, όμως με παρακάλεσε να παρουσιάσω εγώ την εκθεσή της για μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτέ ενέργειας η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των καταναλωτών και η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα πιο δημοκρατικό ενεργειακό σύστημα προ όφελο συνολικά τη κοινωνία. Ενώ θα πρέπει και η συμμετοχή των πολιτών και τη τοπική κοινωνία να αυξηθεί. Ευρύτερα τώρα το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ενεργειακέ τάσει, τι τάσει στην κατανάλωση ενέργεια, δείχνει ότι υπάρχει ε, ψηλό επίπεδο ευσοσύνης, αλλά έλλειψη ανταγωνισμού σε πολλές χώρες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές τιμές ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν έγινε μία δημοσκόπηση, το 30% είπα ότι έχουν πρόβλημα με την ε, εταιρεία παροχής ρεύματος ε, τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να μιλήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο εγώ συγκεκριμένα. Πρέπει να σας πω ότι οι αρχές αγοράς και ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν μια έρευνα για τους παρόχους ενέργειας και ήταν πάρα πολύ καταποτελέσματα. τα αποτελέσματα. Δείξαν ότι πληρώνουν πάνω από 1,2 δις από το 2009 2013 για λογαριασμούς, υπερτιμημένα τιμολόγια και πάνω από τα 2 τρίτα των πελατών δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από πολύ ε, υψηλά και κατάλληλα τιμολόγια. Είχαμε 30% αύξηση των ε, τιμών λιανικής και στη χοντρική είχαμε ρεκόρ αρνητικό πενταετίας. Και κάποιοι χρειάστηκε να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα ζεσταθούν. Στόχο είναι πάντως να δημιουργήσουμε μια ευρύθμως λειτουργού ανταγωνιστική αγορά ενέργεια που θα ωφελεί του καταναλωτέ στόχο είναι ο εκδημοκρατισμό του ενεργειακού συστήματο, βοηθώντα του καταναλωτέ ε, να ιδιοποιηθούν ε, την ενεργειακή μετάβαση, να μπορούν να παράγουν ενέργεια και να είναι ενεργειακώ αποδοτικοί. Θέλουμε λοιπόν ε, να συσχετήσουμε την λιανική και τη χονδρική αγορά καλύτερα και να αντιμετωπίζουμε και τα αίτια της ενεργειακής φτώχειας, προστατεύοντας τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Η έκθεση τονίζει σημαντικές συστάσεις ε, για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αύξηση της διαφάνειας και της αφήνειας ε, στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς, ανάπτυξη κανόνων ε, για σύγκριση στις σελίδες, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να δέχονται προτάσεις για τα πλέον ε, εποφελεί για αυτούς τιμολόγια και θα πρέπει να υπάρχουν, ε, να καταργηθούν τα πρόστιμα για την αλλαγή παρόχων. Αυτό είναι ασύμβατη πρακτική άλλωστε και δεν μπορούν έτσι οι καταναλωτές να αλλάζουν παρόχους ε, και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε συλλογικά προγράμματα μεταγωγής και αλλαγής παρόχων για να μπορούν οι τα κόστη να μειώνονται. Τέλος, η ανάπτυξη της ε, ε, παραγωγής, της ίδιας παραγωγής θα πρέπει να υποστηριχθεί ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως το δικό τους ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψη της Τερέζα η έκθεση να περιοριστεί στην κατανάλωση των οικοκυριών. Πρέπει πια το Κοινοβούλιο να εστιάσει στο ρόλο των πολιτών και στη συμμετοχή τους στην ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, Τερέζα θέλει να ευχαριστήσει του κοιόδης συζητητέ για τη συνεργασία τους και προσβλέπει στην ε, περαιτέρω συνεργασία μαζί τους, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών. Τέλος, η Τερέζα θέλει να προσθέσει ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να εκριζωθεί η ενεργειακή φτώχεια, να προστατεύσουμε από ανταγωνιστικές πρακτικές ε, του ε, σε καταναλωτές, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό απομονωμένοι. Αντίθετα, θα πρέπει να ενωθούμε 28 κράτη-μέλη μαζί, να προστατεύσουμε τους ευάλωτους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε τις αθέμητες πρακτικές. Uh, thank you very much, Αυτά ήταν τα λόγια της εισηγητριάς μας που ακούσατε. Ευχαριστούμε κυρία Γκρίφιν που το παρουσιάσατε. Uh, Πάμε τώρα στις παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών μας που εκπροσωπούν τις πολιτικές ομάδες. Ποιος Λάγκεν από το ΕΛΚ. Äh- Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο δικός μας ο σκιώδης δεν έχει έρθει ακόμα οπότε νομίζω είναι να... καλό είναι να προγραμματίσουμε αρκετό χρόνο για τις προθεσμίες υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό να σας πω τώρα αυτά τα οποία έχει να πει ο κύριος Κέλλη Βεβαίω διάσε την έκθεση και αναρωτήθηκε σε πάρα πολλά σημεία πώς, τι σημαίνει δηλαδή δημοκρατική παροχή ενέργειας πώς οι μεμονωμένες περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να ληφθούν ως μέτρο για προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη και διαπίστωσα πως ε, υπάρχει μία αφελής άποψη για την αγορά ε, ε ενέργεια σε ολόκληρη την ε, έκθεση. Αυτά για εμένα. Τώρα να σου πω την άποψη του συναδέλφου. Τρία πράγματα λέει για τιμές ε, λογαριασμούς και ενεργειακή φτώχεια. Πρώτον, για τις ε, τιμές. Εκεί πέρα η κυρία Γκρίφιν έκανε κάποιες προτάσεις. Ε, λέει ότι θα πρέπει να προσφέρονται μόνο κάποιος περιορισμένος αριθμός τιμολογίων. Κατά την άποψή μου αυτό παραβιάζει την ελευθερία των ε, συμβάσεων και της αγοράς και βέβαια το ότι θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο καταναλωτής στην αγορά. Δηλαδή αν συμμετέχει ενεργά έχει και μία ίδια ευθύνη για την ε, συμμετοχή του ή της. Χρειάζονται λοιπόν ε, κίντρα εντάξει, αλλά αν θέλουν να αλλάξουν τιμολόγιο, αλλά όχι κάποιες διατάξεις δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ποιε θα είναι οι τιμέ στου καταναλωτέ. Αυτό μα λέει η κυρία Κέλλη εδώ πέρα. Για του λογαριασμού τώρα. Συμφωνεί με την ε, εισηγήτρια ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει πολλές άχτες ε, πληροφορίες. Θα πρέπει να είναι απλή ανάγνωση του λογαριασμού και θυμάμαι διαπίστωση του καγκελαρίου του Χέλμουτ Σμιτ του Παλαιού στη Γερμανία που πριν από 25 χρόνια στην πόλη μου στο Αμβούργο είχε πει πως δεν είναι πλέον σε θέση να διαβάσει το λογαριασμό του ρεύματο. Έχει τόσο πολλά πράγματα μέσα που πλέον δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Επίσης, συγκρίσεις ε, και προσφορές ούτε αυτά κολλάνε πάνω σε ένα λογαριασμό όπως προτείνει εδώ πέρα η κυρία Γκρίφιν αλλά δεν ξέρω και οι πλατφόρμες που υπάρχουν που κάνουν αυτές τις συγκρίσεις αν δίνουν αντικειμενικά δεδομένα. Σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αλλάζει κανείς απλά πάροχο αν το θέλει. Αυτά για τους λογαριασμούς. Μετά, ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιθανό ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να το λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο, δύο προτάσεις ακόμα. Δεν γίνεται αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών. Γι' αυτό ο κύριος ε, Κέλλη δεν ε, ε, συμφωνεί με ευρωπαϊκούς ε, δείκτες ενεργειακής στόχιας. Ε, αυτό το οποίο έχει νόημα είναι οι βέλτιστες πρακτικές και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να καλύπτονται οι λογαριασμοί του ρεύματος από τα κοινωνικά κονδύλια. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Παρουσιάστε τις του κ. Το ECR τώρα κυρία Βαν Μπόσιουτς που αντικαθιστά τον κύριο Φόξ. Έχετε το λόγο. Προσωπώ και τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον κύριο Φόξ. Α, τέλειο, λέει ο πρόεδρος. Ακόμα καλύτερα. και θα συνδυάσω τα Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή αγγίζει κάποια κανθόδη θέματα τα οποία πράγματι αφορούν ε, την σημερινή αγορά ενέργειας ε, και η εισηγήτρια δεν διστάζει να θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Έχουμε μια αγορά ενέργειας η οποία έχει πάρα πολλούς φραγμούς και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προστασία των καταναλωτών κτλ. Δυστυχώς, ήθελα να παρατηρήσω πως η εισηγήτρια δεν προτείνει πάντα τις κατάλληλες λύσεις. Η έκθεση έχει ένα ολόκληρο κατάλογο κανόνων ε, που θέλει να επιβληθούν στους ε, παρόχους ενώ ο καταναλωτής θεωρείται ένας παθητικός δέκτης ο οποίος σχεδόν δεν έχει βούληση. Υποτιμάμε νομίζω τον Ευρωπαίο καταναλωτή. δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε νέα διοικητικά βάρη στους ε, παραγωγούς ε, ενέργειας. Επιπλέον ε, διαπιστώνω πως εκεί πέρα που μιλάει για καταναλωτές η έκθεση λέει λίγα πράγματα. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο και με αυτούς αλλά και με τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν θέσεις ε, εργασίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά θα ήθελα να ζητήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος της Άλτε, η κυρία Μλίνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγητή, την εισηγήτρια για την καλή δουλειά της, για την έκθεση και την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ομάδων. Ο ενεργειακός τομέας υφίσταται μια ουσιαστική μετάβαση θεμελιώδη και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν ξεχνάμε το καταναλωτή σε αυτές τις αλλαγές. Μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές είναι σημαντικό ούτω ώστε να αυξηθεί η δύναμη των καταναλωτών και η δυνατότητά τους για πραγματική συμμετοχή όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Ε, και για τους επενδυτές, παραγωγούς και τους εμπλεκόμενους. Όπως είπε η κυρία Γκρίφιν, η έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης για το κόστος και την κατανάλωση καθιστά πολύ δύσκολο για εμάς τους καταναλωτές να σκεφτούμε πραγματικά για τη χρήση της ενέργειας που κάνουμε και να κάνουμε και αλλαγέ στη περιφορά μα. Αν θέλουμε πραγματικά να εμπλέξουμε του καταναλωτέ και να του βοηθήσουμε να μειώσουν και την κατανάλωσή του και το κόστο, το ποσό που πληρώνουν, μέσω του παραδείγματο ε, θα πρέπει να τους δίνουμε ε, προσπελάσιμα ε, στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει το ICT, δηλαδή οι έξυπνοι μετρητέ και γενικά η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τις τιμές χοντρικής και λιανικής. Οι τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνεχώς πέφτουν τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν απεικονίζεται στο, στους λογαριασμούς των καταναλωτών καθώς έχουμε φόρους, ε, τέλη και δαπάνες των δικτύων ε, που βαραίνουν το τιμολόγιο. Για να μεταβούμε επιτυχώς ε, σε μια νέα ενεργειακή οικονομία και να έχουμε μια ευέλικτη αγορά, θα πρέπει να εμπλέξουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της πόλης και τους δήμους και τις κοινότητες δηλαδή, γιατί είναι ο πιο κοντινός σύνδεσμος με τους πολίτες και μπορούν να συνδέσουν την Ενεργειακή Ένωση με τον πολίτη. Ευχαριστώ και ελπίζω να έχουμε και στο μέλλον καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαραγκάλη τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκρίφιν, και την, ε, θέλω να πω και στην ίδια και στην εκπρόσωπό τη, ε, καταρχάς ότι τα, είπανε, τα είπατε πολύ καλά. Ο προσανατολισμός ε, της έκθεσης είναι πολύ καλή. Συμφωνούμε με την θεώρηση, με το όραμα, με τα κριτήρια. Και οι διάφορες απόψεις απεικονίζονται καλά στην έκθεση. Μπορούμε να κάνουμε σημαντικές ε, αλλαγές ε, έτσι στην ε, λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Μπορούμε από το κεντρικό μοντέλο να πάμε σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο. Ε, από, μία, από ένα μοντέλο που ρηπαίνει και που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα να περάσει σε καθαρές μορφές ενέργειας ε, που είναι και ανεξάντλητες. Από, μπορούμε να έχουμε μια πραγματική αγορά με πολλαπλές προσφορές, κάτι που δεν έχουμε και Κυρίως ε, λίγη παραγωγή, ας πούμε, ε, προσφέρουν την ε, ενέργειά τους σε πολλές χώρες. Το ίδιο και διανομής. Επίσης, θα πρέπει οι πολίτες να είναι παραγωγοί και καταναλωτές ταυτόχρονα και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα ελπίζω αγορά μια αγορά με τελικό χρήστη ενημερωμένο, ε, με εξουσία και δύναμη, που μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ε, και δεν θα χαρακτηριζόμαστε. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε online για τις προσφορές, για τις τιμές κτλ. Ε, θα πρέπει να μην χάσει την, ε, το χαρακτήρα της, ε, της να είναι ανοιχτό λέει, στον ιδιωτικό ανταγωνισμό. θα πρέπει να σταματήσουν οι καταχρήσεις. θα πρέπει να άρουμε τα σημαντικά εμπόδια που είναι ουσιαστικά τα ολιγοπόλια, τα οποία κάνουν την μπορούν για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Ε, η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά και αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερασπιστούν οι ίδιοι οι καταναλωτές μια ανοιχτή και δημοκρατική αγορά. Θα εργαστούμε, θα συνεργαστούμε με την κυρία Γκρίφιν και με όλους σας για να συμπληρώσουμε και να κάνουμε πιο συγκεκριμένες τις προτάσεις σας που τις βρίσκουμε σωστές και Θέλουμε να υπάρξει μια ε, ποιοτική αλλαγή και να υπάρξουν πραγματικές ε, νέες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη εξουσία στα χέρια των ε, καταναλωτών και πολιτών μας όλη την Ευρώπη. Από την ΚΟΥΕ. Μπενίτα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη διάθεσή της να συμπεριλάβει και τις προτάσεις μας. η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να περάσει από ένα πιο κεντρικό μοντέλο σε ένα πιο αποκεντρικό και σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, δεύτερη παράγραφο, και σε νομοθετικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν αυτή τη μετάβαση. Ε, παράγραφος 12, εκεί που λέμε για τις, τους φόρους ε, για την ηλιακή ενέργεια. Κάποιες από τις λύσεις βασίζονται μόνο στο να ε, δημιουργήσουμε ένα μοντέλο πιο, πιο ανοιχτό. Όμως ε, θα πρέπει οι πολίτες να ξαναπάρουν τον έλεγχο για να σπάσουν τα μονοπόλια και ολιγοπόλια και να προωθήσουμε και τις ανανεώσιμες ενέργειες. Ε, με προσπάθεια των ε, κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή φτώχεια, πιστεύουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε πολλά. Στην, Ένωση, στην έκθεση θα πρέπει να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα μέτρα, ε, γιατί υπάρχει κοινωνική επιτακτική ανάγκη. Ε, σύμφωνα με τα όσα είπε η ΕΟΚΕ, η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει 50 εκατομμύρια άτομα σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο πιστεύουμε ότι οι εταιρείε δεν θα πρέπει να σταματήσουν να παρέχουν ε, φυσικό αέριο σε οποιονδήποτε λόγω του ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Ε, ειδικά τα φτωχά άτομα, για τα φτωχά άτομα θα πρέπει να έχουμε κοινωνικά τιμολόγια, χαμηλότερες δηλαδή τιμές. για να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική, τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν. Άρθρο 25 ε, της δήλωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ε, γιατί το οποίο λέει, το άρθρο 25, το 25 λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρεπής, ένα σπίτι για όλους τους ανθρώπους, το οποίο θερμαίνεται σωστά κτλ. Ο κ. Σταμπουράνο, από την EFDD Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκρίφιν, που είναι πάρα την απούσα, για τη θαυμάσια έκθεσή της με την οποία γενικά συμφωνούμε. Κυρίως ευχαριστώ ότι έχει ε, και τόσο μακροπρόθεσμη, έτσι, μακροπρόθεσμο όραμα, ας πούμε. Χωρίς ένα τέτοιο όραμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ενέργεια. Επίσης, μαζί σας θα πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρξει αυτή η ενεργειακή μετάβαση, να έχουμε ένα σαφή ορισμό και ενιαίο ορισμό σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο της έννοια του καταναλωτή. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες, ούτως ώστε να μπορούν να προστατεύσουν αυτόνομα αν και πώ θα πάρουν ε, ενεργό ρόλο στην αγορά ενέργειας χωρίς διακρίσεις, ε, χάρη στι ψηφιακέ αρμοδιότητες που θα έχουν, ε, θα πρέπει να γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες, ενημέρωση, γιατί κάτι το οποίο δεν ακούστηκε πολλά σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση είναι το δυναμικό των μηχανισμών που προωθούν την ε, αλλαγή στη συμπεριφορά των ε, καταναλωτών. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά να αξιολογεί και να λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικέ της προτάσεις στην ενεργειακό τομέα. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν φυλάδια ε, τυποποιημένα ε, ενημέρωσης για τα θέματα ενέργειας, εύκολα όμως για τον πολίτη που θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Ιταλία έχουμε πρόβλημα και φαντάζομαι και σε άλλα κράτη μέσα. Και θα πρέπει επίσης οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές ε, με εύκολο τρόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Ακούσαμε ότι υπάρχουν 50, 50 ε, εκατομμύρια άτομα που, έχουν, πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη και αυξάνει αυτό το νούμερο. Δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτούς τους πολίτες πίσω, να τους ξεχάσουμε. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν ένα ελάχιστο ποσό ενέργεια στη διάθεσή τους που θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό αγαθό. Οτιδήποτε αφορά την αυτοπαραγωγή, την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, ε, μια και τον, η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό αγαθό και η σημασία του γίνεται όλο και πιο μεγάλη, αντίστοιχη με του νερού. Ε, και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό αγαθό. Κυρία Σας ευχαριστώ κυρία Κάπελ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Το ενεργειακό σύστημα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν όλο και περισσότερες δυνατότητες οι καταναλωτές να επηρεάσουν την κατανάλωση Τη ενέργειας, εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες και έχουν ξεκάθαρη ιδέα για το από πού θα πρέπει να αγοράζουν την ενέργειά τους. Βεβαίως, κατά την άποψή μας, ε, εδώ πέρα δεν βγαίνουν τα σωστά συμπεράσματα από την κατάσταση γιατί δεν έχουν όλοι οι καταναλωτέ τι ίδιε ανάγκε και επιθυμίες και δεν έχουν όλε οι αγορέ τον ίδιο βαθμό ολοκλήρωση. Και είναι σημαντικό να δοθούν τα σωστά μηνύματα για να δημιουργηθεί μια λιανική αγορά η οποία δεν θα γίνει, δεν θα καθορίζεται από τα κάτω προς τα πάνω αλλά από τον καταναλωτή. Να αφαιρθώ τώρα στα εξή σημεία της ε, έκθεσης. Λοιπόν, για τους παραγωγούς. Ε, δεν πρέπει μόνο οι παραγωγοί να φέρονται σωστά, όλοι συμμετέχονται στην αγορά. Τρίτο ενεργειακό πακέτο. Η αλλαγή ε, παρόχου είναι πάρα πολύ χαμηλή σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες ε, όχι. Το θέμα λοιπόν είναι ο βαθμός του ανταγωνισμού. Διαφάνειας λογαριασμούς. Κοιτάξτε, ακούμε ήδη πως είναι περίπλοκος ο λογαριασμός του ρεύματος και κάποιες χώρες προσπαθούν να επιβάλλουν διαφάνεια, αλλά με κάποια λογική σας παρακαλώ. Το συγκρίσεις δεν έχουν νόημα με άλλους παραγούς πάνω στον ε, λογαριασμό τον ίδιο. Και το ίδιο και με τις ε, φτηνότερες ε, και τυποποιημένες συγκρίσεις. Μην προσπαθούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο, άμα θέλουν συγκρίσει θα κάνουν. Ενεργειακή φτώχεια. Όλοι είναι υπεύθυνοι, όχι μόνο οι πάροχοι και οι παραγωγοί. Είμαστε κατά των ε, επιδοτήσεων, ε, οι οποίες θα επιφέρουν περισσότερου φόρους. Είμαστε υπέρ τη ελάφρυνση από φόρου για να πέσει η τιμή. Και τέλος, κοινωνικό τιμολόγιο, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει καμία δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το πράγμα και έχουμε καταθέσει και τις ανάλογες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε παρέμβαση λοιπόν των σκιωδών εισηγητών και των πολιτικών ομάδων. Τώρα περνάμε στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συνάδελφό μας, ε, την ε, Τερέζα Γκρίφιθ. Υγεία εύχομαι και ελπίζω να αναρρώσει. Είναι ένα θέμα μεγάλης ε, σημασίας γιατί όπως ανέφεραν πολλοί εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων η ανταγωνιστικότητα των τιμών και το γεγονός ότι οι καταναλωτές πρέπει να πληρώνουν την σωστή τιμή είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχει μεγάλη σημασία πώς μπορεί κάποιος να πληρώνει μια τιμή όταν σε όλες τις χώρες έχουμε το ίδιο πρόβλημα δηλαδή μονοπόλιο παρόχου Μπορούν λοιπόν να γίνουν αλλαγές γρήγορα σε άλλους τομείς, αλλά εδώ πέρα είμαστε εξαρτημένοι από τα καλώδια που έρχονται στο σπίτι μας. Τα μονοπόλια λοιπόν καθορίζουν ε, τους λογαριασμούς ε, και αποφάσισαν ότι αυτοί θα φτάσουν πλέον σε δυσθεώρητα ύψη και επιπλέον οι καταναλωτές πληρώνουν τιμές που δεν δικαιολογούνται από τίποτα. Χρειαζόμαστε πραγματικό ανταγωνισμό και κανόνες θα επιτρέπουν στους παρόχους ε, να χρησιμοποιούν τα δίκτυα διανομής για να μειώσουν μέση. Όσον αφορά τώρα την ενεργειακή φτώχεια, είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ριζικής ενεργειακής ε, φτώχειας. Ε, είναι πολυτέλεια για αυτούς ε, το ρεύμα. Καλώς ορίζω λοιπόν την ε, θέληση των πολιτικών ομάδων να καταλήξουμε σε μια καλή εκθέση. Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια προς την ε, εισηγήτρια γιατί έκανε θαυμάσια δουλειά. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν όχι μόνο και καθαρή ενέργεια, βιώσιμη ενέργεια και προσπελάσιμη ενέργεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πρέσιο, ούτω ώστε οι ίδιοι να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν τη δική τους ενέργεια, κάτι που ε, στην χώρα μου δεν διευκολύνεται λόγω των φόρων και να περάσουμε σε μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές ε, ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να συγκρίνουν τιμές, να αλλάζουν εταιρεία γρήγορα, να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους, να κερδίσουν σε ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει, αν θέλουμε να φτιάξουμε την Ενεργειακή Ένωση, χρειαζόμαστε να το κάνουμε συνδέοντας ε, τις ανάγκες των, και βάζοντας ανάγκες των πολιτών στο κέντρο αυτού του εγχειρήματο. Μία αγορά ε, δεν λειτουργεί όταν αποκλεί εκατομμύρια άτομα τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν για να έχουν φως. Ε, η ενεργειακή φτώχεια θα πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα να, να, να ανακόψουμε αυτή την τάση. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να ζούμε στον ίδιο κόσμο, συνάδελφοι. Αλλά αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω σε αυτή την έκθεση ότι υπάρχει κάτι θετικό που μιλάει, και αυτό είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ενεργειακή απόδοση. Αλλά μια και δεν λέμε πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε, είναι σαν να ευχόμαστε να μας την δωρήσει ο Άι Βασίλης. Να σας θυμίσω κάποια πράγματα. Ποια είναι η πιο ε, συγκεντρωμένη, η συγκεντρωτική αγορά στη Γαλλία, στη, ε, στην ενέργεια, στη Γαλλία. Έχουμε μονοπόλια. Ποια είναι η πιο χαμηλή τιμή ενέργειας η γαλλική τιμή, οι γαλλικές τιμές. Σας παρακαλώ λοιπόν, πάψτε πια να μιλάτε για αυτό το γενικευμένο ανταγωνισμό. Όταν έχουμε φυσικά μονοπόλια και για να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η αγορά δεν μπορεί να το οργανώσει καθόλου αυτό το πράγμα, έτσι μακροπρόθεσμα, να οργανώσει αυτό τον ανταγωνισμό. Ε, ο γενικευμένο ανταγωνισμό οδηγεί σε απίστευτη ανασφάλεια. Και τώρα τι θέλετε, ακόμη περισσότερη περισσότερο ανταγωνισμό για να αναστρέψει αυτήν την κατάσταση. Μα τι, τι, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, τι φλήνα θύματα είναι αυτά. Ο Το κείμενο που μας πρότεινε ε, η κυρία Γκρίφιν έχει πολλά θετικά. Η αγορά λιανικής θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφάνεια ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να στηρίζεται σε στέρεε βάσει. Το τρίτο πακέτο, η δημοκρατικοποίηση του ενεργειακού συστήματο, ε, η πρόθεση τη και τη ζήτηση, η καταπολέμηση ενεργειακή φτώχεια, αυτή είναι η φτώχη, οι στόχοι που αναφέρονται από την Τερέζα με μεγάλη σαφήνεια στην πρότασή τη. Είναι σαφέ ότι η συζήτηση για τι ε, αγορέ λιανική δεν μπορεί να ξεχνάει τι τιμέ που προσφέρουν οι αγορέ χοντρικής και θα πρέπει να υπάρχει ε, διαφάνεια, ε, δημοκρατική αγορά και αλληλεγγύη στην αγορά λιανικής. Αυτή είναι η έκκληση που, λέει, που, κάνει η και χαίρομαι γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του τρίτου πακέτου, νομίζω ότι αυτό που αναφέρει παράγραφος 6 για ε, το κόστος, τις τιμέ, ενημέρωση, τιμολόγια είναι βασικό στοιχείο για την, το New Deal και Καταλαβαίνω βεβαίω τι αντιδράσει των operator, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να λογικευτούν και να σκεφτούν ότι έτσι πάει ο κόσμο. Ε, αν θέλουμε να έχουμε ενεργειακή ένωση για το φυσικό αέριο, για την, ε, τον ηλεκτρισμό, για τους μηχανισμούς διακυβέρνησης, ε, θα πρέπει για όλα τα στοιχεία της αγοράς, γιατί να μην ισχύουν και για το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας που είναι η διανομή. Με αυτή τη στιγμή ε, το γεγονός ότι έχουμε ε, διαφορετικά τιμολόγια ε, νομίζω πλήρει το καταναλωτή. Θα πρέπει να πάψει αυτό. Σε ευχαριστώ Ρόιλ. Κοιτάξτε, ε, η έκθεση περιγράφει σωστά το πρόβλημα, αλλά στις λύσεις ε, έχει αστοχήσει λίγο, δοκάρει και έξω. Κοιτάξτε, μιλάτε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει τυποποίηση τιμολογίων, λογαριασμών. Ε, τι, τι τα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω κάθε καταναλωτής μπορεί να λάβει μια απόφαση χωρίς να του την ε, επιβάλλουμε ή υπαγορεύσουμε. Αυτό να το στηρίξουμε, ναι, αλλά δεν ανάγκη να επιβάλλουμε επιπλέον τέλειο, όπως είπαν στην αδελφή. Θεωρώ πως ε, λέτε εδώ πέρα πως θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλλαγή παρόχου. Μα δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Τρίτον, ενεργειακή φτώχεια. Ναι. Τα 5 εκατομμύρια τώρα ε, εγώ θα ε, ήθελα να ξέρω πού τα βρήκατε και ποιοι είναι. Αλλά υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, αλλά η κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι τελείω διαφορετική. Δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και υποθέτω πως μεγάλη ευθύνη για τι τόσο ψηλές τιμές ε, του ρεύματο στην Ευρώπη την φέρουμε εμεί με τις ε, πολλέ μα αποφάσει Και αν λάβουμε πάλι τέτοιε αποφάσει θα γίνει ακόμη πιο ακριβή η ενέργεια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αυτοπεριοριστούμε. Δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται τα πάντα με διάταγμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος τρόπος να καταλήξουμε σε πιο φθηνές ε, τιμές. Και νομίζω πως εδώ πέρα θα βοηθήσει ο ανταγωνισμός και από τη δικιά μου τη χώρα μπορώ να σου πω πως ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος στην αγορά πως ε, το θέμα της αλλαγής παρόχου δεν είναι πλέον ε, κάτι το πάρα πολύ απλό. Και οι εταιρείε οι οποίε κάνουν ό,τι θέλουν του πελάτε ανήκουν σε μια εποχή του μακρινού παρελθόντος. Ευχαριστώ, κυρία Καλά. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο έχω εγώ. και όπου δεν συμφωνώ με τον εισηγητή και αφορά τις έξυπνε ε, τεχνολογίες ε, δεν είναι τόσο αρνητικές μπορούν επίσης ε, να καταστήσουν τους καταναλωτέ πιο ενήμερους και να λειτουργήσει έτσι η αγορά. Και αν λειτουργεί αγορά πέφτουν οι τιμές επίσης. Οπότε νομίζω πως οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να είναι και θετικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Κομισιόν, ο κύριος Διευθυντής. Έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Άκουσα τις ε, συζητήσεις σας και σημειώνω με μεγάλη ικανοποίηση πως ε, σχεδόν όλοι μπορώ να πω συμφωνούμε σε μια θεμελιώδη αρχή. Θέλω να χρησιμοποιήσω την διατύπωση της κυρίας Μούντι. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και εδώ πέρα νομίζω συμφωνούμε είναι μια αγορά ανταγωνιστική που θα λειτουργεί, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτή είναι η αρχή που μας ε, καθοδηγεί. Και κύριε Φεμποσούλ, ναι, ο ορισμός ε, του καταναλωτή πρέπει να είναι ευρύς. Είναι τα νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Όλοι αυτοί είναι καταναλωτές. Λοιπόν, τι όμως ε, λαβαίνουν οι καταναλωτές ε, από την αγορά. Ελάχιστα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για του καταναλωτέ. Αυτό ακριβώ πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα δικαιώματα. Και εδώ πέρα, κύριε Μαγκάλ, χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική προσέγγιση και όχι μια θεωρητική όπω είχαμε μέχρι σήμερα. Να σα ε, εξηγήσω. Υπάρχει σήμερα δυνατότητα να αλλάξει κανεί πάροχο, αλλά καμιά φορά αυτό συνδέεται με ποινέ. Πρέπει να καταργηθούν αυτές απλούστατα. Και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζει κανείς εταιρεία. Μετά, συλλογική αλλαγή παρόχου έχει επίσης ε, βελτιωθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο βεβαίως γιατί πολλοί καταναλωτές μας είναι ισχυρότεροι από μεμονωμένους. Αυξάνεται έτσι η δύναμη των καταναλωτών Τώρα δυναμική τιμολόγηση ή χρέωση μαζί με αυτά τα οποία ακούσαμε από την κυρία Κάλλας και οι έξυπνες τεχνολογίες, ναι, αλλά να μην το επιβάλλουμε στους ε, καταναλωτές, να έχει ο καταναλωτής την επιλογή, αν θέλει να ακολουθήσει δηλαδή μια τυποποιημένη τιμολόγηση, μια δυναμική τιμολόγηση, μπορεί να είναι δική του επιλογή. Μετά οι λογαριασμοί οι ίδιοι, ναι, διαφάνεια. Και σας υπόσχομαι πως θα καταθέσουμε πρόταση ότι η πρώτη σελίδα του λογαριασμού θα πρέπει να είναι παρόμοια σε όλα τα κράτη-μέλη και να περιέχει μόνο τι απαραίτητε πληροφορίε για τον καταναλωτή και όχι όλε αυτέ τι λεπτομέρειε που δεν καταλαβαίνει κανεί. Και κανεί δεν θέλει. Μετά, η σύγκριση των τιμών. Ναι, σημαντικά εργαλεία αυτά και χρειαζόμαστε εδώ πέρα μια πιστοποίηση. Έχουμε πολλά εργαλεία, αλλά καμιά φορά δεν είναι αξιόπιστα και πρέπει να φροντίσουμε να είναι ικανοποιητικά. αυτοπαραγωγή. Ε, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός νομικού πλαισίου αυτή τη στιγμή και πρέπει να τους δώσουμε μια νομική βεβαιότητα για το τι μπορούν να κάνουν και σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το δίκτυο διανομής παραδείγματος χάρη. Μετά, για τα... τις τιμές, τα τιμολόγια. Μιλάτε για τυποποιημένα τιμολόγια. Εδώ πέρα συμφωνώ λίγο με τον κύριο Λάγκεν. Θέλουμε όντως τυποποιημένα τιμολόγια. Αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί όσον αφορά την αλλαγή εταιρεία ε, και δυναμική τιμολόγηση, νομίζω αυτά φτάνουν. Μετά η ανταπόκριση στην ζήτηση και συντομεύω κύριε Πρόεδρε, έξυπνοι μετρητές. Επίσης, οτιδήποτε σχετίζεται με νέα τεχνολογία, δυναμική τιμολόγηση γίνεται μόνο με έξυπνους μετρητές. Επίση αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, αυτό το οποίο είπε η κυρία Μλενέρ, τοπικές ε, δράσεις, ε, τοπικές και περιφερειακές. Ναι, υπάρχουν ενεργειακοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία τέτοια πράγματα. Στη χώρα σας κύριε Πρόεδρε, πήγα ο ίδιος ε, πέρσι σε δύο τέτοια τοπικά περιφερειακά έργα και συνδέουμε τις μονάδες αυτές παραγωγής, όλες ανανεώσιμες επί τη ευκαιρία, βιομάζα, και τέλος η ενεργειακή φτώχεια. Και θα ήθελα να επεκταθώ και στους ε, ευπαθείς καταναλωτές, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Εγώ συμφωνώ με τα μέλη της Επιτροπής που έλεγαν να μην δημιουργηθεί ένα ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δουλειά των κρατών μελών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν ακόμα τέτοια συστήματα να το κάνουν. Και μόλις ε, επέστρεψα από την Σόφια στη Βουλγαρία λοιπόν, η κυβέρνηση προχωράει στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Και ξεκίνησαν πρώτα απ' όλα με το θέμα των εφαθών καταναλωτών και τη ενεργειακή στόχη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είδαμε τις βέλτιστες ε, και τις ορθές πρακτικές άλλων κρατών μελών, τις προσαρμόσαμε στο βουλγαρικό πλαίσιο και θα δείτε το Μάιο θα καταθέσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά μοναδικό και δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών της αλληλοβοήθειας και εδώ πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιτροπές που έχουμε να γίνει αυτό με έναν τρόπο ρυθμισμένο και τακτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι όντως αρμοδιότητα των κρατομέλων, δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μούντι, θα θέλατε να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. καλοδεχούμενε ε, οι παρεμβάσει των συναδέλφων και απαντήσει κομισιών. Τώρα, αυτό που είναι σαφέ είναι ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ενεργειακή φτώχεια, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη συμφωνία για του καταναλωτέ ενέργεια και φαίνεται επίση να υπάρχει συνένεση μεταξύ άλλων και ω προ την ανάγκη ε, πληροφόρησης και διαφάνειας ε, των πληροφοριών για να λειτουργήσει σωστά και μεταξύ άλλων. Επίσης υπάρχει ανάγκη εξέβρεση τεχνολογικών λύσεων. Είπατε ότι απορρίπτει την ιδέα κατά κάποιο τρόπο αυτή η έκθεση. Δεν νομίζω. Είπαμε ε, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες. Και με μια ενωσιακή λύση που θα προωθεί περιφερειακές ε, δράσεις ε, για την ίδια παραγωγή, την αποθήκευση κτλ και τα θέματα της διάνοσης θα πρέπει να τα δούμε. Η Τερέζα νομίζω ότι με πολύ ενδιαφέρον θα μελετήσει όλα τα σχόλια των συναδέλφων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και με τους κοιόδης εισηγητές για να προχωρήσουμε και με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσετε τις ευχές μας και τους στην κυρία Γκρίφιν. Αγαπητοί φίλοι. Η προθεσμή για την κατάθεση τροπολογιών είναι 25 Φεβρουαρίου, ώρα 12 το μεσημέρι. 25 Φεβρουαρίου. Κατάθεση τροπολογιών. Tabling amendments. Thank you very much. Πηγαίνουμε στο σημείο 5. Προς έναν σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση κ. Λάγκεν. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων γίνεται μετά την δημοσίευση τη ε, ανακοίνωση Κομισιόν του Ιουλίου του 2015 για τον ανασχεδιασμό τη αγορά ενέργεια. Μέρο του κ. Λάγκεν περιέχει κάποιε προκατακτικέ απόψει τη Επιτροπή ΙΤΡΕ τι οποίε θα υπόψη του Κοινοβουλίου, προτού δημοσιευθεί η νομοθετική πρόταση τη Κομισιόν στα τέλη του έτου για τον ανασχεδιασμό τη αγορά ενέργεια. Επομένω. Είμαστε μετά τη δημοσίευση τη ανακοίνωση και πριν τη δημοσίευση τη νομοθετική πρόταση από πλευρά Κομισιόν. Ορισμένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι, για παράδειγμα, το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας ε, του εφαρισμού ε, του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ρόλος των επιπτωτήσεων ιδίως για τις μειονονές πηγές ενέργειας και πολλά άλλα θέματα. Προμήθεια φυσικού αερίου. Η Επιτροπή μας θα διεξαγάγει δημόσια ακρόαση για το θέμα στις 17 Μαρτίου. Πολύ σημαντική ακρόαση λοιπόν για τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας τον επόμενο μήνα, σε ένα μήνα από τώρα λίγο πολύ, θα έχουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Όπως βλέπετε, είναι γενικός ο τίτλος της έκθεσης «Ανασχεδισμός αγοράς ενέργειας». Κυρίως όμως αφορά την αγορά ηλεκτρισμού. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του, της, του σε φυσικό αέριο και κάποιοι άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας. Ο κύριος Λάγκεν Παρακαλώ να μας παρουσιάσει τις απόψεις και την έκθεσή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε ήδη τα σημαντικότερα ζητήματα. Ακρόαση στις 17 Μαρτίου και μετά η νομοθετική πρόταση το τέλος του έτους. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα εδώ στον σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς Έχουμε κανονίσει, όπως είπαμε και την ακρόαση, από τις 27 Ιανουαρίου υπάρχει έκθεση μου σε όλες τις γλώσσες. Οπότε, εντάξει, παρουσιάζω σήμερα τα κυριότερα σημεία. Δεν υποθέτω ότι έχουν προλάβει όλοι οι συνάδελφοι είναι την διαβάσουν. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τα βασικότερα σημεία. Θα πρέπει να δοθεί ένα σήμα μήνυμα μέσω των τιμών για τις νέες επενδύσεις. Δεύτερον, να υπάρξει μια νέα προσέγγιση για την ε, ασφάλεια παροχής ε, και το άλλο σημαντικό σημείο είναι η περιφερειακή συνεργασία ειδικά όσον αφορά τις ε, νέες επενδύσεις, ε, διασυνδέσεις και ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με βάση αυτούς τους τρεις στόχους λοιπόν υπέβαλα το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία. Πρώτον, η πρόταση της ε, Κομισιόν όσον αφορά την κινητικότητα των τιμών και των ε, τιμών ε, σε περίπτωση στενοπών στην αγορά που θα πρέπει να δίνουν τα μηνύματα στους καταναλωτές. Επί της αρχής είναι σωστό, εάν καταργηθούν ε, βεβαίως οι ρυθμισμένες τιμές εντελώς δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά υπάρχει εδώ πέρα μια σύγκριση όπως είπαμε μεταξύ των ρυθμισμένων τιμών και των παραπάνω επενδύσεων που ζητάμε. Το άλλο θέμα είναι η ασφάλεια παροχής είναι κατά βάση σήμερα όπως και το ενεργειακό μέγμα υπόθεση των κρατών μελών. Η Κομισιόν θέλει μια νέα ευρωπαϊκή διάσταση χωρίς να υπονομεύει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά θετικά σημεία, τα έχω αναφέρει. Τρίτο θέμα, ενισχυμένη συνεργασία των παρόχων και των παρόχων του δικτύου. Εδώ πέρα υπάρχουν ήδη πάρα πολλά καλά παραδείγματα συνεργασίας. Πολιτικά πρέπει να δούμε αν θα πάμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και αν θα πρέπει να υπάρξει μια επισημοποίηση της συνεργασίας των TSO του δικτύου, των εταιριών δικτύου μεταφοράς δηλαδή. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά μετά όσον αφορά την κατάσταση σε 7 κράτη-μέλη όπου δεν λειτουργεί επαρκώς ο μηχανισμός της ε, αγοράς ε, όσον αφορά τον μετασχηματισμό στις ε, ΑΠΕ και καθώς υπάρχουν εθνικές τρευλώσεις στον ανταγωνισμό και οι αγορές έχουν φτάσει στα όρια τους. Θα πρέπει λοιπόν, προτείνω εγώ, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τρεύλος στον ανταγωνισμό μέσω κρατικών ενισχύσεων και να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές της ε, πολιτικής ανταγωνισμού οι οποίες θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έχουμε την επέκταση του δικτύου και τη μεταφορική ικανότητα μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για μια εσωτερική αγορά ενέργειας, η δικτύωση των κρατών μελών ε, έχει ακόμα μεγάλα κενά, είχαμε μέχρι τώρα στόχο 10% δικτύωσης, τώρα φτάνουμε στο 15%, πρέπει οι να ξεπεραστούν και μετά βεβαίως υπάρχει το θέμα της τιμολόγησης η οποία θα αντικατοπτρίζει την, ε, το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Το θέμα λοιπόν των ΑΠΕ μετά. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια παραδείγματα όπως στη δική μου τη χώρα πως η μόνιμη επιδότηση με σταθερές τιμές εγγυημένες πλέον δεν ε, ανταποκρίνεται στην κατάσταση των ε, γερών και οπωσδήποτε δεν είναι ανταγωνισμός να έχουμε εγγυημένες τιμές για 20 χρόνια. Οπωσδήποτε απαιτείται η μετάβαση στη ΑΠΕ αλλά θα πρέπει να γίνει με βάση την αγορά και πρέπει να ενισχυθεί και η αγορά intraday. Μετά όσον αφορά τους, ε, τις εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο διανομής. Είχαμε το πρώτο ενεργειακό πακέτο και τώρα έχουμε περαιτέρω προτές για κάτω των 100.000 χρηστών όπου θα πρέπει να υπάρξει μια αποδέσμευση ε, του δικτύου. Αυτό το θεωρώ λάθος ε, γιατί υπάρχει ζήτημα διαθεσιμότητας προσωπικών δεδομένων που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταία μου παρατήρησε όπως όλες οι εκθέσεις έτσι και αυτή έχει κάποιο όριο λέξεων ε, και θα ήθελα να ληφθεί αυτό υπόψη από τους συναδέλφους όταν θα κρίνουν την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, Κύριο Ζανατό, δύο λεπτά ο καθένας. Τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε γίνεται. Όχι, όχι, θα έρθει ο Επίτροπος, λέει ο Πρόεδρος. Το σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου Λάγκεν είναι μία βάση αφετηρίας. Υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει όμως να διερευνηθούν περαιτέρω. Πολύ σύντομα. Για το επιστημιολογικό κομμάτι. Η βασική επιστημολογία δεν βασίζεται στην ε, διείδηση των ενεργειακών ε, επιχειρήσεων. Ε, συνεχώς γίνονται κλήσεις ε, για να ασχοληθούμε με τους κοινούς στόχους από κοινού αλλά θα πρέπει ε, να ξεπεράσουμε τα, εθνικά προνόμια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω, δεν έχω σε καμία περίπτωση διάθεση να αμφισβητήσω το ρόλο των κρατών μελών και την αρμοδιότητά τους για να καθορίσουν το ενεργειακό μείγμα. Αλλά εδώ περνάμε κάτι, μιλάμε για κάτι πέρα από το ενεργειακό μείγμα που έχει και επιπτώσεις ε, στο, στο ενεργειακό, στο κλιματικό συγγνώμη, θεματολόγιο. Το να ανασχηματίσουμε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει καταρχά να ενσωματώσουμε τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ε, το κείμενο του Ντλάγκεν εδώ μιλάει να φτάσουμε στο 30%. Αλλά πώς θα φτάσουμε στο 30% εάν πρώτον δεν υπάρχει καμία υποστήριξη ε, μέσω προγραμμάτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Δεύτερον, 19. Ε, εάν βάλουμε και τον το οικονομικό στοιχείο, ε, αντισταθμιστικά ωφέλη στους operator. Παράγραφος 23. Τρίτον, υποθέτουμε στην παράγραφο 20 ε, μιλάμε για τις διάφορες προτεραιότητες χωρίς να αναφέρουμε καθόλου ε, την αποθήκευση των, ε, της ενέργειας. Ε, χωρίς να εξασφαλίσουμε αυτά τα τέσσερα στοιχεία δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το 30%. επίση. θα πρέπει ε, συνέχεια να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες οι οποίες ε, πηγαίνουν από τα κράτη-μέλη στην Ένωση ε, με σεβασμό την αρχή της επικουρικότητας και στον ενεργειακό τομέα και όσο μπορούμε θα πρέπει να δίνουμε κοινέ απαντήσεις. Αυτό, σημαίνει, αυτό ισχύει και για την, το σχεδιασμό της, της αγοράς. Αλλά το κείμενο του Λάγκεν ε, μιλάει κυρίως για εθνικές λύσεις ε, και εθνικές στρατηγικές. Νομίζω ότι κινείται εδώ προς λάθος κατεύθυνση και δίνει εξουσίες σε πολυμερή φόρουμ και όχι ε, σε μια διαδρομή που θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος. οι επαγγελματίες χρήστες καναλωτές. Ε, είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση τη Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω και εγώ δύο λόγια. Θέλω να τονίσω τρία σημεία. Η έκθεση γενικά μου φαίνεται ισορροπημένη. Και θα τη στηρίξουμε. Να τονίσω λοιπόν τρία σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Πρώτον, το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα. Ο εισηγητής ε, είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στο μέλλον να υπάρχουν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Δεύτερη ιδέα, αυτό που μόλις ακούσαμε, ανώνυμες πηγές ενέργειας να είναι πιο πολύ προσανατολισμένοι στην αγορά. Συμφωνούμε. Τρίτο σημαντικό στοιχείο, η περιφερειακή πτυχή των αγορών ενέργειας για να έχουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Δηλαδή τους ίδιους κανόνες για όλους. Και είναι και οι κανόνες που βλέπουμε στην τριπτές μέτρων για την ενέργεια. Αυτό είναι τα θετικά. Έχω και τρεις ε, κριτικές. Το πρώτο δεν βλέπουμε το ρόλο των συμβολίων ή συμβάσεων μακράς διάρκειας. Δεύτερον, αρνητική προσέγγιση σε σχέση με τις αγορές ισχύω power markets που είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της ενέργειας. Και τρίτο στοιχείο που λείπει από αυτήν την έκθεση είναι μια διαφοροποίηση μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Δεν έχει αξιολογηθεί το κόστος της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ήταν και σύντομος. Εκ μέρους της Άλτε, ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ, η συνάδελφος ε, έμεινε στην Πράγα. Θα σας πω εγώ τις παρατηρήσεις που θα έλεγε. Να ευχαριστήσουμε βέβαια τον εισηγητή κύριο Λάγκεν. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού είναι σημαντική για να έχουμε ασφάλεια φοδιασμού και για περιορισμό των εισαγωγών από τρίτες χώρες και μείωση του κόστου ενέργειας και για τους ιδιώτες και για τις επιχειρήσεις, μείωση εξάρτησης. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση, είναι σημαντικό να παραμείνουμε, να έχουμε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στόχους, πρέπει να επιτευχθούν ε, σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος, πρέπει να είναι προβλέψιμο και σταθερό το ρυθμιστικό περιβάλλον που θα σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Ταυτόχρονα η Ένωση θα μπορέσει να φέρει ε, σε πέρα σε αυτές τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις ε, με ε, τη μεταρρύθμιση του ETS και με την έρευνα και την ανταμοιβή, την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πολιτικών, χωρίς όμως ε, αυτό να γίνει σε βάρος α, τρίτων άσχετων περιοχών που θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό της αγοράς. Και θα, πρέπει να δούμε και αυτή την ιδέα περί αγορών ισχύω. Επίσης ε, η πρόταση Λάγκεν μας βρίσκει σύμφωνος, ε, δηλαδή ότι πριν ρύθμιση των τιμών θα πρέπει να γίνουν πιλωτικά σχέδια γιατί υπάρχουν διάφοροι συμβαλόμενοι που ε, θα ήθελαν κάτι αντίστοιχο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο αξιόπιστο τέτοιο παράδειγμα στις ευρωπαϊκές αγορές. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ εκ μέρους των κύριο Στούρμες, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι στην έκθεση αυτή ε, πολλά είναι αυτά που μας βρίσκουν σύμφωνος. Πρώτα απ' όλα η σχετικά επιφυλακτική προσέγγιση απέναντι στις ε, εθνικές πληρωμές National Capacity Payments. Πολλές φορές ασκούνται πιέσεις από ολιγοπόλια και δεν είναι και εύκολο να καταλάβει κανείς ε, τους λόγους γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Κύριε Λάγκεν, Είστε υπέρ, λέτε, της περιφερειακής συνεργασίας, αλλά μετά λέτε ότι ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για το σκοπό αυτό. Όμως ο κ. Ζανονάτο με βρίσκει πιο σύμφωνος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τις που κάνει για την αγορά φυσικού αερίου, ε, γιατί εκεί πιστεύω ότι βλέπουμε πού πρέπει να οδεύσουμε και με την αγορά ηλεκτρισμού. Αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τα περιφερειακά ωφέλη, μάλλον τα ωφέλη της περιφερειακής συνεργασίας, χρειάζεται αυτή η διακυβέρνηση. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να διατυπωθεί κάπως καλύτερα ή πιο φιλόδοξα αυτό το σημείο. Αυτό που μου λείπουν για το ETS λέτε ότι πρέπει να ενισχυθεί. Δεν κάνετε όμως προτάσεις συγκεκριμένε. Ίσως όταν δευτερολογήσετε θα μπορούσατε να μου απαντήσετε με ποια συγκεκριμένα μέτρα προβλέπετε την ενίσχυση του ETS. Επίσης, η ανταπόκριση στη ζήτηση. Είναι ίσως ο πιο φθηνός τρόπος για να έχουμε ευελιξία και στις περιφερειακές αγορές, άρα πρέπει να τονίσουμε αυτό το σκέλος. Και τέλος, ε, η ιδέα σας είναι κάπως κατά των ανάσων πηγών ενέργειας. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχει αυτή η τάση στην έκθεση για να είναι πιο ισορροπημένη. Όσο οι αγορές βλέπουμε να έχουν τόσες πολλές αστοχίες ε, στον τομέα του άνθρωπου κτλ. Χρειαζόμαστε ε, να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές, να στηρίξουν τις ανανεώσιμες. Κυρία Ένστα από την ΚΟΕ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θεωρώ πως ε, είναι θετικό το ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον ανακοινώνται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δηλαδή στο μελλοντικό πλαίσιο, μια περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά το δίκτυο αλλά δεν προχωράμε όσο πρέπει. Σημαντικό σημείο είναι το σημείο 26 με το ενεργειακό μείγμα και η αγαπημένη σας εκεί πέρα πυρηνική ενέργεια. Αυτό το θεωρώ λάθος και δεν πρέπει να γράφουμε τέτοια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να φύγει. Σημαντικό και σωστό είναι η κριτική τοποθέτηση για τον μηχανισμό δυναμικότητας ε, των δικτύων, όπως επίσης και τα μηνύματα για την ε, τιμολόγηση. Βεβαίως είμαστε σαφώς κατά αυτών των εθνικών μηχανισμών ε, δυναμικότητας, αφενός γιατί δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο με βάση το οποίο θα μπορούσε να γίνει και βεβαίω σημαίνει πως θα υπήρχε μια σημαντική αλλαγή της αγοράς την οποία είχαμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη και νομίζω πως ε, συνεισφέρει περισσότερο σε μια περιχαράκωση και όχι σε μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και θα πρέπει να υπάρχει και μια αξιολόγηση αντικτύπων για τέτοια πράγματα και να είναι πιο έντονες οι διατυπώσεις όσον αφορά την επιφυλακτικότητα απέναντι στην ε, αγορά αυτή που φτάνει στα όρια της. Σας ευχαριστώ Ταμπουράνο για το EFTD. Ευχαριστώ τον κύριο Συγητή Έχει πολλά θετικά στοιχεία. μα αρέσει η κριτική στο μηχανισμό δυναμικού, όπω και οι προλαλήσαντε. Θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση τη ενεργειακή αγορά θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο κλειδί για να περάσουμε πιο γρήγορα σε μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές ε, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των στόχων κλίματο και ενέργεια. Ε, εμείς με ποια λογική θα σα πω θα κάνουμε τις τροπολογίε τροπολογίες μας. Οι ανανεώσιμες θα πρέπει να μπουν στο κέντρο να δούμε πώς θα συμμετάσχουν ε, στο δίκτυο και τι σχήματα σταθερά υποστήριξης θα έχουν. Ελπίζω να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να αναγνωρίσουμε και τον ρόλο του παραγωγού καταναλωτή. Κάποιε διαστάσει τη αγορά θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη, γιατί η αγορά δεν είναι ένα απλό μηχανισμό διαμόρφωση των τιμών. Και απαιτεί όχι μόνο πληροφορίε λεπτομερεί ε, των φορέων για εξωτερικά στοιχεία θα πρέπει να είναι και στοιχείο συμμετοχής, εμπλοκής διαφόρων φορέων. Όλα τα μοντέλα αγοράς είναι καλά ε, με, δια, με κειμενόμενες τιμές. Υπό τον όρο όμως ότι θα υπάρχουν ε, εγγυήσει ότι θα αποκλειστεί κανένας. Οι διακοιμάσεις να μην οθήσει εκτός αγοράς κανέναν Ευρωπαίο πολίτη. Με ειδική προσοχή στους πιο ευπαθείς. Αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτηση τα 50 εκατομμύρια πολιτών στην Ευρώπη που βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια, το 10% δηλαδή, του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Εάν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα πράγματα, για ποια ενεργειακή ένωση μιλάμε πάντα για το θέμα της συμμετοχής. Θα πρέπει να έχουμε εργαλεία οικονομικά για να αυξήσουμε τον αριθμό παραγωγών ε, παύλα καταναλωτών. Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι γίνονται ε, μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα 20-30 χρόνων. Και με αυτόν τον τρόπο ε, βοηθούν και βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς. Σήμερα είμαστε σε μια φάση επιδοτήσεων κτλ που έδωσαν την προτεραιότητα σε κάποιους τομείς και ε, υποτίμησαν κάποιους άλλους. Θα πρέπει, μην ξεχνάτε, ότι η αγορά θα πρέπει να δημιουργεί αντισταθμιστικά συστήματα, ούτω ώστε όλοι οι φορείς να ανταγωνίζονται οι μεν τους δε ε, ισότιμα, ας πούμε. Αν μιλάμε για φιλελεύθερη αγορά, θα πρέπει να αφορά όλους αυτή η αγορά. Κυρία Κάπελ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση που μας δείχνει την αναγκαιότητα για μια νέα αγορά ενέργειας και μας λέει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να είναι βιώσιμη αυτή η αγορά. Να αναφέρω όμως κάποια θεμελιώδη πράγματα για εμένα. Έχουμε την αυστριακογερμανική τιμή τιμολογίων που θα πρέπει νομίζω να διατηρηθεί γιατί αλλιώς θα υπάρχει μεγάλο χώρος για την χώρα μου κατόπιν θα πρέπει να είναι ίση η όρη του ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς ενέργειας και παρόχους φυσικού αερίου. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί βεβαίως δεν αφορά μόνο την ολοκλήρωση της αγοράς ε, χοντρικής και μεγάλων πελατών αλλά και την λιανική. Η ασφάλεια παροχής και του στήματος θα πρέπει να ενισχυθεί και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν με τρόπο γρήγορο, άμεσο θα έλεγα και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τις ε, στενοπούς και την διαχείρισή τους. Όσον αφορά τώρα το πριμ ε, δυνατότητας μεταφοράς για διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ καλός ορισμός των νέων εταιριών και βέβαιως για το ποιος επομίζεται το κόστος για τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα το συνολικό κόστος θα πρέπει βεβαίως να συμπεριλαμβάνεται στην ε, τιμή. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για όλους συμμετέχοντες στην αγορά και να υπάρχει διαφάνεια, παραδείγματο χάρη μέσω και καθημερινών προκηρύξεων, αλλά βεβαίως ε, και θετικά και αρνητικά δικαιώματα όσον αφορά τους ε, πρωτογενείς παραγωγούς. Τέλος θα πρέπει οι διαγωνισμοί να γίνονται μέσω μιας ηλεκτρονικής ε, πλατφόρμας και βεβαίως να δούμε το τι θα γίνει με την ε, αγορά και τους ε, ενδιάμεσους και την, τον έλεγχο της αγοράς μέσω τηλεκατεύθυνσης. Θα πρέπει επίσης λοιπόν να υπάρξουν νέα ενεργειακά προϊόντα και οι ρυθμιστές θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους και οδησίγητες. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους. Έχω πάρα πολύ μεγάλο κατάλογο. Ένα λεπτό ο καθένας δυστυχώς. Μπλάνκο Λόπες πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στη Δημιουργία ε, διασυνδεδεμένης αγοράς ηλεκτρισμού με πυλώνα, ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές, ε, εφοδιασμό σε ενέργεια για να μπορούμε να έχουμε και προστεστιμές και εξασφαλισμένη παροχή ηλεκτρισμού. Βέβαια θα πρέπει να αυξηθούν οι διασυνδέσεις στην εσωτερική αγορά για να πάψουμε να έχουμε ενεργειακές νησίδες όπως είναι η Βυρική Χερσόνησος. Επίσης, αυτοί οι μηχανισμοί δυναμικότητας, αυτές οι αγορές δυναμικότητας είναι σύμπτωμα του προβλήματος που είναι η έλλειψη ενοποίησης, ολοκλήρωσης που υπονομεύει την ασφάλεια εφοδιασμού. Όμως το κλειδί σε αυτό το νέο σχεδιασμό είναι η αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης, η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, διαχείριση της ζήτησης, ανανόσιμες πηγές ενέργειας και η ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι οι πολίτες ή επίσης ε, και η ανάπτυξη ευφυών δικτύων με επίκεντρο η νέα αγορά ε, ενέργειας να έχει τον πολίτη και να μην αποκλείεται κανείς. Πρόεδρος, One να σας πω ότι την επόμενη μία ώρα και 30 λεπτά έχουμε συνάντηση με τον Επιτρόπο Αρίας Κανιέτη και έχουμε παρόμοιο θέμα ε, οπότε μπορείτε και εκεί να θέσετε τα ερωτήματά σας. Έχουμε και στις 17 Μαρτίου την ακρόαση, όπως σας είπα, που πάλι θα έχει το ίδιο θέμα. Επόμενος ο ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω, να δούμε την ενεργειακή ροή από βορρά προς νότον, ειδικά στη Γερμανία όπου έχουμε ενεργειακή ροή από δυσμάς προς Ανατολάς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την ε, νέα πραγματικότητα των τιμών χωρίς να σταματάμε σε εθνικά σύνορα. Το στόχος δικτύωσης 15% είναι πάρα πολύ σωστός κατά την ε, άποψή μου. Βεβαίως είναι ζήτημα σχεδιασμού και υπάρχει και ζήτημα αγορών ε, όταν φτάνουν αυτές τα όρια τους με δημόσιους διαγωνισμούς και με τους κανόνες που ισχύουν για τα χρηματιστήρια που θα πρέπει βεβαίως ε, πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν ε, μόνο τις πραγματικές συναλλαγές των εταιριών και να μην αποτελέσουν ένα νέο αντικείμενο κερδοσκοπίες για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλέπουμε παραδείγματο χάρη και θα πρέπει να δώσουμε βάρος όπως στη Βουλγαρία να καλύπτεται το κόστος ε, της παραγωγής και να μην πωλείται το ρεύμα σε τιμή κάτω του κόστου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πολύ ο συντονισμός, ε, η ενοποίηση είναι λέξεις κλειδιά για μια νέα αγορά ενέργειας ε, και ο ρόλος της διεύθυνσης είναι πολύ σημαντικός. Ε, ο εισηγητής δεν έχει κάνει μια πολύ φιλόδοξη έκθεση παρόλα αυτά, υπογραμμίζει απλά το ρόλο του Άσερ ως οργανισμού συνεργασίας των θεστικών αρχών. Συμφωνώ με τον κύριο Τούρμες ότι θα πρέπει να δούμε ε, τι δυνατότητε που πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη, αλλά να δώσουμε και μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση. Οι ανανοσπιστέ πρέπει να ενταχθούν στην αγορά, η παραγωγή, η ολική, η ηλιακή πρέπει επίσης να ενταχθούν, αλλά να κάνουμε και ένα βήμα πιο πέρα και θα κάνω σχετικές προτάσεις. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος που δίνεται ε, στα εφή δίκτυα και στις διασυνδέσεις. Αυτό είναι σημαντικό πραγματικά για την αγορά Ναι, Κυρία Νίμπλερ, επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συντομότατα θα ήθελα να πω πως είναι πάρα πολύ καλή έκθεση του κυρίου Λάγκεν. Θέτει τα σωστά ερωτήματα, αγγίζει τα σωστά θέματα, κάνει τη σωστή πολιτική αξιολόγηση. Το σημείο 26 εμένα δεν με ενοχλεί. Το σημείο 26 θεωρώ πως είναι σωστό, λέμε πως θέλουμε μια ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι σωστό. Επίσης το ενεργειακό μείγμα είναι υπόθεση των κρατών μελών. Αυτό το γράφουν οι συνθήκες και αναλόγως πρέπει να κινηθούμε. Δεύτερον, θεωρώ πως είναι σωστά αυτά τα οποία λέει για τις αγορές που είναι στο όριο. Πράγματι θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες αγορές, αλλά Βεβαίως ε, θα πρέπει να δεχτούμε αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα ο εισηγητής ε, στη μεταβατική περίοδο, αλλά θα πρέπει η Κομισιό να τα δει λεπτομέρως. Και τρίτο, η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εδώ πέρα συμφωνώ με τον κύριο Λάγκεν πρέπει να κατευθύνουμε την αγορά μέσω των κατάλληλων μήνυματων. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή ε, είναι πολύ συνενετική. Κάποιε ρωτήσαν τον κύριο Λάγκεν. Στο σημείο ε λέτε ότι το δυναμικό, το εθνικό, οι εθνικές αγορές δυναμικού ε, καθιστά πολύ δύσκολη την ενσωμάτωση, την ενοποίηση της ε, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντιβαίνει στην ενεργειακή πολιτική. Δεν συμβαίνει το αντίθετο. Για να έχουμε μια καλή αλυσίδα θα πρέπει καταρχά να έχουμε εθνικό δυναμικό. Πώ θέλετε να φτιάξετε αυτή την αλυσίδα και να είναι αν δεν βασιστούμε στην, στο εθνικό δυναμικό. Επίση, ε, δεν θέλετε σταθερέ τιμέ, ε, επιδοτήσει, ε, προτεραιότητα στην πρόσβαση, προνόμια των κρατών πολύ ωραία. Αλλά χάρη σε αυτά μπορούμε εμεί να σα δίνουμε, χάρη σε αυτά τα προνόμια, εμεί στη Γαλλία, α πούμε, μπορούμε να σα δίνουμε ενέργεια και εσεί να μα δίνετε εμά. Ε, με μια καλή συμπληρωματικότητα. Παράλληλα, θέλετε και ένα ε, κανονιστικό πλαίσιο. Δεν αντιβαίνει αυτό όσα λέτε. Και στο σημείο 2, στο σημείο 5 μάλλον, κάνετε, θέλετε κάποιες, ε, κάποια κίνητρα. Πετε μου τελικά, θέλετε απελευθερωμένη αγορά, είτε το αντίθετο. Δεν θέλετε να... Δεν μπορούμε να έχουμε και ελευθερία και ταυτόχρονα αριθμιζόμενη αγορά. Κύριε Συγητή, να προσθέσω δύο πράγματα. Καταρχά, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ασυντόνιστα, ασυντόνιστες ροές στο δίκτυο. Δεύτερον, έχουμε ε, μεγάλη εξάρτηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εξωτερικούς ε, προμηθευτές, κυρίως κράτη. Πρέπει να στηριχθούμε και στις ανανεώσιμες. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια μελέτη και να αναλύσει μια νέα αγορά ηλεκτρικού που να, είναι, που να δίνει ε, προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και να ε, παρεμποδίσει τις διαρροές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ο κ. Μπόλχαρτ, ο Διευθυντής, εκπρο... εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ξανά εγώ. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πρόεδρε, κάνετε μία εισαγωγή και μιλήσατε για την συνδιασύνδεση της αγοράς χοντρικής και με τις αγορές ε, λιανικής. Το συζητήσαμε στην έκθεση Γκρίφη. Στη συζήτηση ακούσαμε για την ευπάθεια των καταναλωτών, ε, για τη ζήτηση της ενέργειας. Όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε, παρότι σωστά ε, επιλέξατε να κάνετε δύο διαφορετικές εκθέσεις για τα δύο θέματα αυτά. Εδώ μιλάμε για την αγορά χοντρικής. Τι παίζετε εδώ. Υπάρχει συνένεση καταρχά μεταξύ τη Επιτροπή και τη Κομισιόν ότι χρειαζόμαστε ανοιχτέ και ενοποιημένες αγορές που θα δίνουν ασφαλή ε, προσιτή ενέργεια, βιώσιμη ενέργεια, ε, με σεβασμό των κλιματικών στόχων. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μαζί. Και νομίζω το γενικό στόχο όλοι το συμμερίζονται. Τώρα να τονίσω κάποια από τα σημεία τα οποία ε, συζητήθηκαν εδώ και που αφορούν το σχεδιασμό της αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια χοντρικής. Καταρχάς, να αναφέρω το, ε, το σύστημα ε, διαμόρφωσης των τιμών. Στην έκθεση Λάγκεν υπάρχει υποστήριξη για ειδικέ τιμές σε περίπτωση έλλειψης. Και επίσης μας ζητάει να υπάρχει μια περίοδος δοκιμής. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορείτε να βασιστείτε μόνο στις τιμές ε, έλλειψης. Καταλαβαίνω βέβαια ε, την ανησυχία που υπάρχει πίσω από αυτό το σημείο και θα πρέπει τουλάχιστον εδώ να προβλέψουμε μία αναθεώρηση μετά από ένα διάστημα για να δούμε τι εμπειρία έχουμε αποκομίσει. Να πω γενικά, κάτι που σκέφτηκα όταν διάβασα την έκθεση και που το είπε η κυρία Νίμπλε. Είναι μία έκθεση που αφορά, ε, που θέτει τα σωστά ερωτήματα, δίνει σε, μεγάλο βαθμό καλές απαντήσεις και μας βάζει και σε σκέψη. Εσείς, Πρόεδρε, τώρα θέσατε το θέμα των, της, του που κολλάει η ροή της, της ενέργειας. Θα το κοιτάξουμε εμείς ως Κομισιόν Έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας. Βλέπω ότι το αφεντικό μου έφτασε, ο Επίτροπος ο κ. Κανιέτε, γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσω. Έγινε μια συζήτηση για την περιφερειακή συνεργασία. Δεν υπάρχει ομοφωνία εδώ. Η έκθεση Λάγκεν δεν μιλάει τόσο πολύ για την... δεν τονίζει πολύ τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας. Ο κύριος Τέρμες και ο κύριος Τσορίνο ε, μίλησαν για την ενίσχυση των ε, αρμοδιοτήτων Acer. Είναι σημαντική η περιφερειακή συνεργασία και αν θέλετε δεν έχετε άλλη επιλογή από το να έρθουν, να πιο κοντά οι διάφοροι operators, οι TSO. Κάτι άλλο που λέει πολύ σωστά και ε, παρουσιάζει πολύ σωστά η έκθεση Λάγκεν είναι ο μηχανισμός οικοδόμησης δυναμικού. Ε, ο κ. Σταμπουράνο και ο κ. Τέρμες υποστηρίζουν αυτό το σημείο. Εμείς δεν είμαστε κατά τέτοιων μηχανισμών, αλλά θα πρέπει να αποδείξετε καταρχήν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για αυτό το δυναμικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια περιφερειακή παραγωγή ε, που αφορά ε, όλη την περιφέρεια και όχι μόνο το κράτος μέλος. Γιατί μπορεί οι γείτονέ σου να έχουν ε, υπερβάλλον δυναμικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που χρειάζεται, εκεί που υπάρχει ανάγκη. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε, και το λέει και η έκθεση Λάγκεν, είναι να αποφύγουμε τις τρευλώσεις της αγοράς. Και τέλος, μια και ακούστηκε και αυτό, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πέρα από το σχεδιασμό της αγοράς, θα έχουμε και ρυθμίσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού, Κανονισμό για την ετοιμότητα απέναντι στο κίνδυνο, που μοιάζει λιγάκι ως νομοθετική πρόταση, και θα σας τα πει ο κύριος Κανιέτε, ε, μα, την πρόταση που έχουμε στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, θέλουμε και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα να έχουμε αντίστοιχε προτάσει, ούτω ώστε η ασφάλεια ανεφοδιασμού να αντιμετωπίζεται σε περιφερειακό επίπεδο με όλα τα κατάλληλα εργαλεία που θα σας παρουσιάσει ο Επίτροπος. Ευχαριστούμε και καλωσορίζω τον Επίτροπο Κανιέντε, αλλά θα ήθελα πρώτα ο εισηγητής μας, ο κ. Λάγκεν, να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους, κυρίως τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, μου είχαν στείλει κάποια πράγματα εκ των προτέρων. Δεύτερον, να αναφερθώ σε κάποια πραγματάκια που θα τα ακούσουμε και στην ακρόαση. Ο πρώτος είναι ο ρόλος της ΕΣΑ. Σε αντίθεση με τα όσα ακούστηκαν, εγώ έδωσα και παραδείγματα. Μιλάω για διασυνοριακές αρμοδιότητες σε διασυνοριακές περιπτώσεις και να υπάρχει είτε ισοδυναμία συστημάτων καθώς επίσης και στην έγκριση ε, των αδειών. Μιλάμε λοιπόν για συγκεκριμένη επέκταση της αρμοδιότητας ε, και βεβαίως το δεύτερον οπωσδήποτε υποστηρίζω το στόχο της Κομισιόν να ενσωματώσει τις ανανεώσιμες φυγές ενέργειας πλήρως στην αγορά. Και άρα η πρόταση μείωσης ε, των επιδοτήσεων δεν περιορίζεται μόνο στις ανανεώσιμες αλλά ακριβώς και στην πυρηνική ενέργεια βλέπουμε πως η Κομισιόν ε, με διαστόματος ε, του Επιτρόπου Ανταγωνισμού Αλμούνια μιλάει για 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να δοθούν ε, σε νέο πυρνικό εργοστάσιο στη Μεγάλη Βρετανία και το ενέκρινε αυτό και θεωρεί πως δεν υπάρχει καμία στρέβλωση του ανταγωνισμού. Νομίζω πως έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πάρα πολύ και για την στήριξή σας. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ όλους τους ε, σκιοδησηγητές, όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Να σας πω πως οι προθεσμοι για είναι 21 21η Μαρτίου το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Για μένα αυτό σημαίνει μεσάνυχτα, ε. και 59 το βράδυ, λοιπόν, 21 Μαρτίου. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαιρόμαστε που είστε πάλι εδώ. Έχουμε έναν δομημένο διάλογο, κοινοβούλιο με την Κομισιόν και παρουσίαση του πακέτου του αερίου ε, από τον κύριο Κανιέτε, τον Επίτροπο Κλίματος ε, και Ενέργειας. Όπως ίσως ε, θυμάστε, στις 16 Φεβρουαρίου 2016 η Κομισιόν ενέκρινε το λεγόμενο πακέτο του αερίου που περιέχει δύο νομοθετικές προτάσεις για την ασφάλεια παροχής αερίου και διακυβερνητικές συμφωνίες με, τρεις χώρες, με τρίτες χώρες και δύο μη νομοθετικές ε, προτάσεις, στρατηγική θέρμανσης και ψήξης, ε, LNG και αποθήκευση φυσικού αερίου. Δύο προτάσεις λοιπόν πολύ σημαντικές ε, από την σκοπιά της ενεργειακής αγοράς. Κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ να παρουσιάσετε λοιπόν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρουσιάσω το πακέτο ασφάλεια ενεφοδιασμού στην Επιτροπή σα. Όταν ήρθα εδώ πριν από ένα χρόνο για να παρουσιάσω τη Στρατηγική Ενεργειακή Ένωση, Σα υποσχέθηκα ότι θα επανέλθω και κάθε φορά που θα έχουν προτάσει θα σα τι παρουσιάζω. Φυσικά θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλέ προτάσει στο χρονοδιάγραμμά μας, θα, θα έχετε πολλέ ευκαιρίε να με ξαναδείτε. Ε, σήμερα είμαι εδώ για να παρουσιάσω αυτό το ουσιαστικό πακέτο ασφάλιση ανεφοδιασμού. Πριν πω στι λεπτομέρειε, θα ήθελα να περάσω σε κάποιε ερωτήσει που έχετε θέσει τι πρόσφατε εβδομάδε. Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το πακέτο και γιατί το χρειαζόμαστε τώρα. Απλά χρειαζόμαστε αυτό το πακέτο γιατί είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και πολύ ε, ευάλωτοι στι ενεργειακέ ελλείψει. Χάρη στον κανονισμό του 2010 για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την πρόοδο στι διασυνδέσει, ε, του κανόνε ε, για τα δίκτυα και την αντιστροφή του, της ροής του αερίου. Αποφύγαμε την κρίση, μια κρίση κλίμακας ε, όπως το 2006 και το 2009. Αλλά η κατάσταση είναι ακόμα προβληματική ε, και οι δοκιμές αντοχής έδειξαν ότι είμαστε πολύ ε, ευπαθείς σε πολλές διαταραχές στην ασφάλεια, στον εφοδιασμό του φυσικού αερίου. Ε, πάνω από το μισό της ενέργειάς μας πρέπει να το εισάγουμε. Πολλές χώρες εξαρτώνται από έναν προμηθευτή ε, και όλα αυτά ε, συμβαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ε, απρόβλεπτου γεωπολιτικού κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε τώρα για να αποφύγουμε νέα κρίση. Και αυτό ισχύει και για την ενεργειακή μετάβαση και για την μετάβαση σε εκπομπές με μειωμένες, μειωμένες διοξείδιο του άνθρακα. Η μόλυνση του φυσικού αερίου, από, η μόλυνση που προκαλεί το φυσικό αέριο είναι η μισή από τον άνθρακα ε, και είναι πολύ σημαντικό για να ε, στηρίζει και την παραγωγή μας σε αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Ε, πρέπει να πω όμως ότι η στρατηγική μας δεν είναι να, παρουσια, να να χρησιμοποιούμε περισσότερο αέριο, αλλά να το χρησιμοποιούμε πιο ε, έξυπνα. Ε, και να χρησιμοποιούμε την ενέργειά μας πιο αποτελεσματικά. Για κάθε ε, αύξηση κατά 1% της ενεργειακής αποδοτικότητας, οι εισαγωγές του ε, φυσικού αερίου πέφτουν κατά 2,6%. γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή αποδοτικότητα θα είναι προτεραιότητα στην Ενεργειακή Ένωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος για τη μετάβαση και στο μεταξύ θα πρέπει τα σπίτια μας να θερμάνονται και οι οικονομίες μας να χρησιμοποιούν την ενέργεια με βιώσιμο και ασφαλή τρόπο. Ε, αυτό ήταν για το ε, πώς. Τώρα ε, ήταν για το γιατί. Τώρα θα σα μιλήσω για το πώ. Έχουμε δύο νομοθετικέ προτάσει στο πακέτο μα, ε, που είναι συμπληρωματικέ και δύο στρατηγικέ που θα ήθελα να συζητήσουμε. Καταρχά να ξεκινήσω με την πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ασφάλειας του εφοδιασμού. Ε, οι δοκιμέ αντοχή του 2014 μας έδειξαν κάποιες βασικές και πικρές αλήθειες. Έδειξαν ότι οι εθνικές πολιτικές ανέργειας δεν βοηθάνε για την ασφάλεια των εφοδιασμού των γειτόνων. Οι εξωτερικές απειλές ε, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνου και τα εμπορικά συμβόλαια εφοδιασμού δεν είναι αρκετά διαφανή για να εντοπίσουμε οποιοδήποτε κινδύνο στον εφοδιασμό. Όλα αυτά τα σημεία ε, δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη συνεργασία και γι' αυτό τι προτάσει μα εστιάζουμε στο συντονισμό και στην αλληλεγγύη. Οι προτάσει μα θα εξασφαλίσουν ότι όλε οι χώρε θα έχουν ε, θα δίνουν αρκετή ενέργεια στα νοικοκυριά και στι κοινωνικέ υπηρεσίε σε περίπτωση κρίση. Αυτό σημαίνει ότι θα προστατεύουμε περισσότερο του μη προστατευόμενου καταναλωτέ στι γειτονικέ χώρε σε σχέση με του δικού μα. Ένα, μια προβλητική δράση και ένα σχέδιο κατεπίγουσας ανάγκης, θα, αυτά θα γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο και θα αξιολογούμε και τους κινδύνους. Ε, επίσης προτείνουμε ε, μία α, αυτόματη κοινοποίηση στα συμβόλαια αερίου τα οποία διαρκούν πάνω από 1% σε περίπτωση που το μερίδιο της αγοράς από τον προμηθευτή είναι πάνω από το 40% στην αγορά συνολικά. Πολλοί θεωρούν, ανησυχούν γι' αυτό, γιατί πιστεύουν ότι οι Βρυξέλλε θα έχουν τη μύτη του σε εμπορικέ συμφωνίε. Αλλά δεν πρόκειται να κατασκοπεύουμε, απλώ θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ε, σε κάθε περιοχή για, την, ε, για τον εφαδιασμό σε φυσικό αέριο. Ε, αυτό θα μα βοηθήσει να εντοπίσουμε τι περιπτώσει όπου χρειάζεται ε, αξιολόγηση κινδύνου και προληπτικά μέτρα ε, και πρέπει να τα προσαρμόσουμε μάλιστα αυτά. Α περάσουμε τώρα στι ε, διακυβερνητικέ συμφωνίε. Ε, μερικοί από εσά θα ρωτάτε γιατί θέλετε να αναθεωρήσουμε μια νέα νομοθεσία. Ξέρω ότι ο κύριος Καρίνς, ο κύριος Τικαστήλιο Βέρα και ο κύριος Γιούρκ δουλεύουν ε, ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα των ε, συμφωνιών. Ε, δείχνει, αυτό δείχνει πόσο φρέσκια είναι η νομοθεσία μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι συμφωνίες αυτές δεν συμμορφώνονται με το ε, νοσιακό δίκαιο της πολιτικές. Όταν ε, υπογραφεί μια συμφωνία δεν μπορεί να ξανανοίξει και οποιασδήποτε νομικές διαδικασίες δεν μπορούν να διορθώσουν την ε, ζημιά που μία ε, ασύμβατη διακυβερνητική συμφωνία έχει στην ασφάλεια ανεφοδιασμού. Όταν σκεφτείτε ότι το 1 τρίτο από τι 124 ε, διακυβερνητικέ συμφωνίε έχουν διατάξει που δεν συμμορφώνονται με το νοσιακό δίκαιο, βλέπετε πόσο προβληματικέ ε, μπορεί να είναι. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε μια ε, υποχρεωτική αξιολόγηση οποιασδήποτε συμφωνία πριν υπογραφεί. Η Κομισιόν θα κοινοποιήσει το κράτο μέλο ε, για οποιαδήποτε ε, αμφιβολίε μέσα σε έξι εβδομάδε και θα δώσει μια τελική γνωμοδότηση για συμβατότητα συμβατοτητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσα σε 12 εβδομάδε. δηλαδή, απλά καμία χώρα δεν πρέπει να υπογράψει μια συμφωνία μέχρι να δώσει τη γνώμη τη Κομισιόν και θα πρέπει να τη λάβει εν συνεχεία το κράτο μέλο υπόψη αυτή τη γνώμη. Ε, εάν παρόλα αυτά υπογράψει τη συμφωνία παρά την ε, αντίθετη γνώμη τη Κομισιόν, εμεί θα ε, προσφύγουμε εναντίον αυτού του κράτου. Ε, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι αυτοτιμωρία. Θα, είναι είναι ένα διάλογο ανάμεσα στην Κομισιόν και στο κράτο μέλο με βάση τα στοιχεία και την ανάλυση για την επίπτωση τη ε, διακυβερνητική συμφωνία. Ο στόχο είναι απλό. Να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι συμφωνίε δεν έχουν αρνητική επίπτωση στην ενεργειακή ασφάλεια της ε, Ευρώπης και στη σωστή λειτουργία της εσωτερική αγοράς. Είναι οι δύο νομοθετικές προτάσει αυτέ που προτείναμε την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στι δύο στρατηγικέ. Καταρχάς, ε, το LNG, ε, στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και στρατηγική αποθήκευση. Ε, η, ο ανεφοδιασμό LNG ε, αυξάνεται και αυτό θα βοηθήσει την ε, αντοχή μας ε, θα έχουμε περισσότερε πηγέ ανεφοδιασμού και θα μειωθούν οι τιμέ. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να συνδεθεί η Ευρώπη με τι αγορέ LNG ε, χάρη στην κατάλληλη υποδομή. Έχουμε ε, σημαντικό δυναμικό επαναεριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και μπορούμε να εισάγουμε LNG κυρίω από τι ΗΠΑ, Αλγερία, Νιγηρία, Κατάρ κτλ. Αλλά το βασικό, ε, οι βασικές υποδομές βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη. Σε άλλε περιοχέ Ευρώπη. ε, ε οι υποδομές δεν είναι ικανοποιητικές. Γι' αυτό θα πρέπει στα, στη Βαλτική, στην Κεντρική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Νοτιοδυτική Ευρώπη να αυξήσουμε, αυξήσουμε τις υποδομές. Θα πρέπει ε, η, η συμφόρηση η, να, να έρθει ε, θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πηγές ανεφοδιασμού, ε, να υπάρχει ανταγωνισμό στις τιμές σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να υποφεληθούμε από τις διεθνείς αγορές LNG. Μέχρι στιγμής ε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο με τους διεθνούς μας εταίρους, ούτως ώστε να έχουμε ελεύθερες, ρευστές και διαφανείς αγορές. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την η Ιαπωνέζικη Προεδρία του G7 να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με την Αυστραλία και να έχουμε διαλόγους υψηλού επίπεδου με την Αλγερία, Καναδά και Ηνωμένε Πολιτείες. Και να ολοκληρώσω εκεί από όπου ξεκίνησα. Δεν μιλάμε μόνο για περισσότερο αέριο. Ε, μην ξεχνάμε ότι ο τομέα τη ε, θέρμανση και τη ψήξη ε, καταναλώνει το τη μισή μα ενέργεια και τα τρία τέταρτα του φυσικού μας αερίου και είναι από τις πιο αναποτελεσματικές στην οικονομία μας. Το 60% των παλιών κτηρίων έχουν παλιούς καυστήρες και έχουν χαμηλά, ε, χαμηλούς συντελεστές απο, ενεργειακής αποδοτικότητας. Έχουμε χαμηλά επίπεδα ανακαίνιση των κτηρίων και βλέπετε ότι έχουμε τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Η στατική μας εστιάζει στην άση των φραγμών για την ε, μείωση των εκπομπών από τα κτίρια και τη βιομηχανία. Θα πρέπει ε, να συνδέσουμε τις, τα δίκτυα ε, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώσουμε το κόστος για το καταναλωτών και να εξασφαλίσουμε την αποθήκευση ε, των ανανεώσιμων που είναι πιο φθηνές. Ε, επίσης θα πρέπει τα ποσοστά ανακαίνησης να ε, επιταχυνθούν. Θα πρέπει ε, οι αναποτελεσματικοί καυστήρε σε πολυκατοικίε να αντικατασταθούν. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε και τις κατάλληλες επιλογές ε, και να χρησιμοποιήσουμε ε, τα εργαλεία που έχουμε, όπω το ΕΦΣΥ. Στο ΕΦΣΥ, χάρη στο ΕΦΣΥ έχουμε επενδύσει σε project ανακαίνησης, ανεδιακή ανακαίνησης, σε πολυκατοικίε στη Γαλλία, που μειώνει την κατανάλωση ενέργεια σε αυτά τα κτίρια κατά 75% και μειώνει το λογαριασμό για περισσότερα από 40.000 σπίτια. Αλλά ε, χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα από αυτά. Ε, το Smart Finance for, small, for Smart Buildings είναι μια ε, καινοτομία που θα διευκολύνει την πρόσβαση ε, σε νέους και καινοτόμους ε, μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης για ανακαινήσεις που σκοπό έχουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το σημερινό πακέτο θέλει να εξασφαλίσει ασφάλεια, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας και συνεχεία θέλω να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο και κυρίως με την Επιτροπή σας, ούτω ώστε αυτές οι προτάσεις να γίνουν νομοθεσία. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η δέσμη μέτρων για όλους μας. Υπογραμμίσατε και εσείς τη σύντομη ομιλία σας τα πιο σημαντικά στοιχεία, πόσο σημαντικό είναι το υγραέριο, οι λύσεις επίσης που είπατε για 36 χώρες, άρα δεν αφορούν μόνο εμάς αλλά και οι γειτονικέ μας χώρες, τις χώρες ενεργειακής κοινότητας. Μιλήσατε νομίζω και για συλλογική αγορά φυσικού Για πρώτη φορά το είδαμε σαν επίσημο γραφό της Κομισιόν να αναφέρεται ρητός ως επιλογή. Πρόληψη κρίσεων. Εξίσου σημαντική με την επίλυση κρίσεων. Άρα πρέπει να προλαμβάνουμε τις κρίσεις και επίσης το σημαντικότερο, κοινοτική προσέγγιση. Γιατί σίγουρα μπορεί να υπάρξει από μία χώρα κρίση σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό, αλλά δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα του εφοδιασμού μόνο μία χώρα, εφόσον προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Για αυτό είναι και σημαντική κοινοτική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα έρχομαι στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Και δίνω καταρχά τον λόγο εκ μέρου έλεξη τον κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο γιατί βεβαίως η πρωτοβουλία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά εισάγει ενέργεια κάθε χρόνο 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι γίνεται και ποιες ε, τιμές είναι ανεκτές. Βλέπουμε πως στον Βορρά υπάρχουν αρκετά μεγάλες δυνατότητες διαθέσιμες. Η Νορβηγία, παραδείγματο χάρη, ή στον Νότο, στην Αδριατική, στην Κύπρο. Έχουμε πολλές ε, δυνατότητες στον τομέα του φυσικού αερίου να αναπτύξουμε τις δικές μας ε, πήγες και αυτό νομίζω πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Τώρα όσον αφορά το κλίμα, η μετάβαση από τον άνθρακα στο αέριο θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλες εξοικονομήσεις εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε όλα τα σχετικά έργα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται σε μια θέση ανταγωνιστική όσον αφορά και τις ε, τιμές της ε, ενέργειας. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, είναι σημαντικό το σχέδιο Juncker και για αυτές τις δυνατότητες των δικτύων μαζί με το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη γιατί βεβαίως γνωρίζουμε πως ε, βασικό πρόβλημα είναι και τα θέματα των ε, υποδομών. Γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς το θέμα της αποδίκευσης ε, να προωθηθεί γιατί θα μας ε, βοηθήσει πάρα πολύ και η μετάβαση εξαρτάται και από τη δυνατότητα αποθήκευσης και από τη δυνατότητα της δικής μας παραγωγής βεβαίω. Σας ευχαριστώ. Νταν Νίκα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γεια σας κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε την υπόσχεσή σας και σας ευχαριστώ που έρχεστε εδώ να μα παρουσιάσετε κάθε νομοθετική δέσμη μέτρων, η συγκεκριμένη που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντική, διότι αφενό μα δίνει τη δυνατότητα πετύχουμε έναν πολύ σημαντικό στόχο, 30% ανανόσιμες πηγές ενέργεια. Νομίζω είναι εφικτό με τα μέτρα που μα προτείνατε σήμερα, γιατί χωρί μια στρατηγική για το φυσικό αέριο είναι σχεδόν ανέφικτη η στρατηγική αυτή γιατί δεν έχουμε μια ε, εναλλακτική δυνατότητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους μας για τις εκπομπές εξιδίου του άνθρακα. Εξίσου σωτική σημασία είναι η διασύνδεση μεταξύ όλων των πηγών ε, και παρόχων φυσικού αερίου. Για όσους δεν το κατάλαβαν, πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο που αγοράζουμε ε, το φυσικό αέριο, από που έρχεται. Αλλιώς ε, δεν έχουμε την ε, δέουσα ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση τώρα σε αυτό το φυσικό αέριο. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά κάποιος έχει το θάρρος να θέσει το ζήτημα αυτό, που είναι πρώτα και πάνω απ' όλα πολιτικής φύσεως ξέρετε τι συνέβη κάποιο χειμώνα με το φυσικό αέριο και γενικώ ε, ε, τα, τα σημεία ε, σύνδεσης θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη δυνατότητα μεταφοράς. Μιλήσατε και για περιφερειακή συνεργασία. Πώς θα λειτουργήσει και τι ποινές προβλέπονται για μη συμμορφούμενα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διοργανικές συμφωνίες. Υπάρχει στο Συμβουλίο Πλειοψηφία για τις ε, εξάντε τιμές. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ξέρω ότι υπήρξαν αντιρρήσεις προς αυτή την προσέγγιση. Τέλος, όταν εγκριθεί αυτή η δέσμη, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος. Αναφερθήκατε και εσείς στον τομέα της μεταφοράς, των μεταφορών. Δεν θα πρέπει να δούμε και την είσοδο του φυσικού αερίου στον τομέα της ναυσιπλοείας. Καζανεύσκη, Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση προς τον Επίτροπο. Στο πλαίσιο του πακέτου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πετύχει και τον έλεγχο των εμπορικών συμβάσεων. Σε σχέση με την ε, ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο μηχανισμός ελέγχου, πώς ακριβώς τον έχετε φανταστεί και τι είδους κυρώσεις, τι είδους ποινές θα επιβάλλονται. σε πρώτος παράσταση αυτής της αρχής περί ασφάλισης αποδιασμού. Αν δηλαδή αποφανθεί σχετικά η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο Κλοντ Τούρμες, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με κάτι που ελπίζω να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στρατηγική θέρμανσης και ψήξης. προσυπογράφω σχεδόν όλα τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό. Αλλά νομίζω ότι χάνεται την ευρύτερη εικόνα, κύριε Επίτροπε, για ε, να έχουμε πραγματικά επενδύσεις στην θέρμανση και ψήξη. Έχουμε τώρα ένα περιβάλλον με χαμηλές ε, τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πώς λοιπόν μπορούμε να ταγωνιστούμε. σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό το οποίο λείπει εντελώ από τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γιατί είναι τόσο χαμηλέ οι τιμέ πετρελαίου, θα παραμείνουν τόσο χαμηλέ και αν ναι, είναι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν οικονομικέ γεωπολιτικέ πτυχέ. Και νομίζω ότι όλοι οι ειδικοί για την ενέργεια ε, τους τελευταίους τρεις μήνες μιλάνε για ακριβώς το θέμα αυτό, τις χαμηλές τιμές πετρελαίου και τις επιπτώσεις του. Και δεν, κάνει, δεν λέει λέξη όμως η Κομισιόν για αυτά τα θέματα με αυτό το έγγραφο. Σας παρακαλώ λοιπόν πείτε μας κάτι παραπάνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Εμείς οι πράσινοι θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, ε, εξάντε μέτρα. Σας ε, ε, συμφωνούμε με την προσέγγισή σας, αλλά σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να έχουμε μια καλή στρατηγική γιατί πολλά κράτη-μέλη έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να θέλουν να παραμείνουν στο στενό αυστηρό εθνικό σχεδιασμό. Υπάρχουν κάποια σενάρια για το φυσικό αέριο και αυτά, σε αυτά βασίζεται τη στρατηγική σας. Η κατανάλωση φυσικού αερίου μειώνεται στην Ευρώπη ήδη. Γιατί να ανεβεί στα κτίρια. δεν βλέπω ε, μια τέτοια τάση και μιλάτε, ε, λέτε, θα μειώνεται το φυσικό αέριο κατά 2,6 προσθέσουμε για μία ε, ποσοστία μονάδα αύξηση. Στη βιομηχανία είναι λίγο πολύ σταθερά τα πράγματα, στι μεταφορέ. Εντάξει, είπατε για την αυσιπλοή, αλλά δεν είναι και πολύ σημαντικά τα ποσοστά. Και μας μένει ηλεκτρική ενέργεια. Με το ETS ελπίζουμε κάποια στιγμή να ε, αποδώσει. Εγώ Νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη στρατηγική σε σχέση με τον άνθρακα. Αλλά επειδή αυτές οι μονάδες φυσικού αερίου δεν θα λειτουργούν για χιλιάδες ώρες, αφισβητώ την μελέτη αντικτύπου. Ναι. Βλέπετε τι λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι τεράστια ευθύνη της Κομισιόν. Λέτε θα έχουμε τόση ε, χρήση φυσικού αέριο στην Ευρώπη. Τι θα γίνει με τις επενδύσεις, μήπως θα τις πληρώσουν στο τέλος οι καταναλωτές. Μην είμαστε υπεραισιόδοξοι λοιπόν σε αυτά τα σενάρια του φυσικού αέριο. Κύριε Επίτροπε, έχετε οποιαδήποτε απάντηση στις κριτικές και επιφυλάξεις για αυτά τα σενάρια για το φυσικό αέριο. Τέλος. Ο ελέφαντας, ε, μέσα στην δεν τον βλέπει κανένας. Nord Stream. Κόβεται ο πρόεδρος, κόβει τον ομιλητή. Όχι, θα την τελειώσω την πρόταση. Προτείνεται να γίνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων στο υγραέριο, αλλά δεν λέτε ούτε μια λέξη για το τι θα γίνει με το Nord Stream. Διακόπτεται, μιλάνε ταυτόχρονα οι δύο. Κύριο Σιλικιώτη παρακαλώ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχο για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Η στροφή τη ένωση προς το ευρωπημένο φυσικό αέριο αποτελεί αναφίβολα μια θετική εξέλιξη γιατί πρώτα θα επιτύχουμε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και θα μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση από τους αγωγούς και θα δημιουργήσει μια ευέλικτη ενεργειακή αγορά. Εν τούτης, για να επιτύχουμε πραγματικά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, είναι σημαντικό οι τερματικοί σταθμοί υγροποίησης να αξιοποιούν και τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Ε, κάνατε αναφορά στην εισαγωγική σας παρέμβαση ότι Κατά κανόνα εισάγουμε σήμερα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατά, την Αργερία. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι στην ανακοίνωση της Κομισιόν για τη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο επιβεβαιώνεται πως η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί μια υπεσχόμενη μελλοντική πηγή ενεργειακού εφοδιασμού για την Ένωση. Ε, λόγω και των κοιτασμάτων ενό κράτου μέλου τη Κύπρου αλλά και τη ευρύτερη περιοχή, ωστόσο απουσιάζει από την ανακοίνωση μια ολοκληρωμένη πρόταση για αξιοποίηση των προοπτικών που υπάρχουν στην περιοχή. Ε, για παράδειγμα θα μπορούσε η Ένωση να στηρίξει τη δημιουργία ενό θερματικού υγροποίηση ε, στην Κύπρο συμβάλλοντα έτσι καθοριστικό στη μείωση τη ενεργειακή εξάρτηση τη Ένωση, αλλά και στην ενίσχυση τη ενεργειακή τροφοδοσία της. Ε, ένα τέτοιο έργο θα μείωνε βεβαίω και τι περιφερειακέ ανισότητε όσον αφορά την πρόσβαση στο γροπημένο φυσικό αέριο, στόχο που έχει τεθεί ω προτεραιότητα τη Κομισιού, γιατί ξέρουμε ότι στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη υπάρχει σοβαρή ε, κενό στην ενεργειακή ασφάλεια. Όσον αφορά την ανακοίνωση και αναφερθήκατε και στην εισαγωγή σα για τι διακυβερνητικέ συμφωνίε, έχουμε έντονου προβληματισμού κύριε Επιτροπέ καθώς μετατρέπει τα κράτη σε ενεργειακά εξαρτημένα ποιόνια της Κομισιό. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να πετύχει η Κομισιό εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχο και αξιολόγηση όλων των διακυβερνητικό συμφωνιών. Δεν γίνεται να μην επιτρέπεται στα κράτη να συνάπτουν μια διακυβερνητική συμφωνία αν δεν δοθεί πρώτα έγκριση από την Κομισιό, τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακή ασφάλεια. Τα μέτρα αυτά υπονομεύουν κατά την άποψή μα την εθνική κυριαρχία, εκμηδενίζουν την εθνική ευελιξία και εμποδίζουν τα κράτη από το να συνάπτουν πολυεπίπεδε και πολυδιάστατε συμφωνίε βάσει των συμφερόντων λαών. Επίση, αγνοούν και ακυρώνουν τι εθνικέ ενεργειακέ ανάγκε στην περιφέρεια με κίνδυνο να κυριαρχήσουν έτσι τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιριών και τα συμφέροντα των ιδιωτών. Πώ μπορεί η Κομισιόν να ζητά τέτοιε εξουσίε όταν η ίδια αποδέχεται πω ο κανονισμό που μόλις πριν λίγες μέρες έχει ανακοινώσει για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και αναφερθήκατε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη λόγω της ενεργειακής απομόνωσης. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται ρητά ότι ο καλισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο και στη Μάλτα. Άρα θεωρούμε ότι Thank από τη στιγμή που υπαρχουν ενα απομενωμένα κράτη-μέλη ε, δεν είναι σωστό να πάρει αυτές τις υπερεξουσίες Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε το ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε σήμερα για ποιο λόγο είναι απαραίτητο το πακέτο του αερίου για το 2016 και ποιες είναι οι προτάσεις εφαρμογής του. Είναι σημαντικό αυτό και τονίσατε ότι πάνω από 50% του αερίου στην Ευρώπη εισάγεται και πως κάποια κράτη-μέλη είναι εξαρτημένα μέχρι και 70% από έναν προμηθευτή. Και είπατε πόσο σημαντικό είναι το αέριο για, την... για το να φύγει η οικονομία μας από τον ε, άνθρακα. Είπατε παραδείγματο χάρη πως 1% μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα σημαίνει 6% λιγότερες αγωγέ φυσικού αερίου. Επίσης είπατε πως ακόμα και αν επιτύχει τους ε, στόχους της για το κλίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται περισσότερες υποδομές ε, φυσικού αερίου. Γιατί μειώνεται η ευρωπαϊκή παραγωγή, αυξάνονται οι εισαγωγές LNG. Χρειάζονται λοιπόν νέοι τερματικοί σταθμοί και έχουμε κάποια συγκέντρωση κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και ότι το αέριο είναι πάρα πολύ σημαντικό ως ε, καύσιμο ανάγκης για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Άρα το ερώτημά μου. Πώς θα στηρίξει η Κομισιόν το να έχουμε σταθμούς ε, αερίου οι οποίοι θα είναι ανταγωνιστικοί που θα χτιστούν από ιδιώτες, από ιδιωτικές επιχειρήσεις για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, για να είναι φτηνή η ενέργεια. Και δύο ερωτήσεις για την ψήξη θέρμανση που αναφέρατε και είναι βεβαίως ε, σημαντική. τι ρόλο αποδίδεται στο φυσικό αέριο, ειδικά όσον αφορά την ελαστικότητα της αγοράς ενέργειας για την οποία μιλήσαμε ε, σήμερα. Δηλαδή να πάμε σε κοινή παραγωγή και τηλεθέρμανση ή βιοκαύσιμα. Ποια απάντηση έχουμε όσον αφορά το να γίνει το σύστημα και οι αγορές ενέργειας πιο ευέλικτες και ελαστικές και δεύτερον ποιες ε, προτάσεις έχετε όσον αφορά τον ε, συνδυασμό και τη σύνδεση της αγοράς τηλεθέρμανσης με την αγορά ηλεκτρισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Αγαπητοί συντονιστές. Λοιπόν, απαντήστε τις ερωτήσεις ε, των συντονιστών και μετά στους υπόλοιπους ε, κύριε Επίτροπε. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συντονιστές. Ο κύριος Ρούμπιχ είπε πως ε, είχαμε την δυνατότητα τοπικής παραγωγής η Νορβηγία είναι πράγματι πολύ αξιόπιστος πάροχος αλλά έχουμε και τα νέα ευρήματα στην Μεσόγειο στην ε, Κύπρο, στην Αίγυπτο, εκεί στα, στα διάφορα πεδία εξόρυξης ε, του Λεβάντε όπως λέγονται. Λοιπόν, για την ανάπτυξη τώρα του στρατηγικής του LNG υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη το πρώτο είναι δάνεια, το δεύτερο είναι επιχορηγήσεις. Πρέπει να τα συνδυάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά όταν χρηματοδοτούμε κάποια έργα. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν με την στρατηγική αυτή του LNG και το πώς θέλουμε να σχεδιάσουμε την αγορά είναι να έχουμε πιο στοχευμένα έργα και να είναι κυρίως έργα κοινού συμφέροντος. Να εστιάσουμε δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά για να έχουμε μια διασυνδεδεμένη και ευέλικτη αγορά. Και είπατε και κάτι άλλο σημαντικό. Οι γραφειοκρατικές ε, καθυστερήσεις με αυτές προβλέπονται σε οποιοδήποτε έργο. Είχαμε 10 χρόνια ε, ε, όταν είχαμε τον κανονισμό των ευρωπαϊκών δικτύων. Τώρα είναι στα 4 χρόνια. παρόλα αυτά. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα γιατί είναι σοβαρό το πρόβλημα. Μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση χρηματοδότησης, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονται χρόνια. Και βεβαίω η Κομισιόν εργάζεται με ομάδες ε, υψηλού πολιτικού επίπεδου για να δοθεί πολιτική στήριξη σε έργα μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου στη Βαλτική, στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη και αλλού. Και λειτουργεί αυτό γιατί όταν έχει τον Πρωθυπουργό ε, και δίνει πολιτική στήριξη βεβαίω, ναι. Μετά έχουμε τοπικέ περιφερειακέ αρχές και όλα αυτά τα πράγματα. Α δούμε, ας δούμε τον νότιο διάδρομο. Από το Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα, ε, λύσαμε τα προβλήματα και έχουμε μόνο ένα ζήτημα εκεί που βγαίνει ε, ο που καταλήγει ο διάδρομος στην Ιταλία, στην Πούλια. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Μετά. Αν σας αλφό σας επέμεινε στην περιφερειακή συνεργασία. Οπωσδήποτε είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ποιος ε, είναι ο στόχος ε, αυτού του πράγματος που κάνουμε για την ε, ασφάλεια παροχής ενέργειας. Είναι μια ολιστική προσέγγιση. Λέμε μέχρι 31 Μαρτίου 2017 κάθε κράτος μέλος να μας πει ποιοι είναι οι προστατευμένοι πελάτες. Αυτό είναι εθνική απόφαση. Η κάθε χώρα λέει ότι έχω αυτούς τους ε, προστατευμένους ε, πελάτες ε, και έχω κάποιες προδιαγραφές αλλά πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι αυτοί. Το Νοέμβριο λοιπόν 2018 Ο Έντσο λοιπόν θα πρέπει να καταρτήσει και τα σχετικά σενάρια για να ξέρουμε τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά όμως οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Και αυτή η αξιολόγηση είναι κάτι το διαδικό θα έλεγα, γιατί κάθε κράτος μέλος πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση, αλλά μετά σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και μετά όλα αυτά θα πρέπει να έχουν κάποια προληπτικά σχέδια, σχέδια ανάγκης που θα εγκριθούν μέχρι 1η Μαρτίου 2018. Εμείς έχουμε υποβάλει κάποια πρότυπα για να έχουν όλα τα σχέδια την ίδια λογική. Θα αξιολογήσουμε αυτά τα σχέδια, αλλά βεβαίως ε, Αυτά αφορούν ε, τις καταστάσεις ανάγκης. Υπό κάπα λειτουργεί η αγορά. Να συντονιστούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λύσουμε τυχόν προβλήματα. Γιατί βλέπετε ότι ένα, ένα κράτος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί ένα κράτος να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μόνο του και εκεί πέρα απαιτείται αλληλεγγύη. Γεγονός είναι πως η απομάκρυνση των μεταφορών από τον άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό ακριβώς αύριο έχουμε μια κοινή συνάντηση με τους ε, αντιπρόεδρους Κατάινεν και Σεύκοβιτς για το πώς ε, όλοι οι αρμόδιοι επίτροποι θα δουν το θέμα αυτό ε, στις μεταφορές τις οδικές και τις θαλάσσιες. Και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έρχομαι άρα στο ερώτημα του κυρίου Τούρμες που είναι το δύσκολο. Αν δηλαδή η Κομισιόν υπερτιμά την ζήτηση του αερίου. Κοιτάξτε, η πρότασή μας βασίζεται σε κάποια σενάρια που είναι, είναι προβολές, δεν είναι προβλέψεις, είναι διαφορετικό αυτό. τα σενάρια αξιολογούν το τι αντίκτυπο θα έχουν τα μέτρα της πολιτικής και το σενάριο αναφοράς με βάση τις τωρινές τάσεις μας δείχνει το τι θα συμβεί αν συνεχίσουν να ακολουθούν τη διαπολιτική τα κράτη-μέλη να γίνει τίποτα άλλο. Και λέμε Εντάξει, μπορεί να είμαστε μεταξύ 380 και 550 PCM μέχρι το 2030, αλλά θα συζητήσουμε δύο σημαντικές πολιτικές εδώ μέσα. Τις ανανεώσιμες, τη σχετική οδηγία, την οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας και να δούμε μετά τι επίπεδο ενεργειακής αποτελεσματικότητας θέλουμε. Αυτά όμως ε, κυμαίνονται, δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διαβεβαίωση. Ακολουθούμε μία πορεία λοιπόν τα σταδιακής από τον άνθρακα, αλλά έχουμε ένα επίπεδο ενεργειακής αποτελεσματικότητας το οποίο θα αποδεχτούμε εμείς και τα κράτη-μέλη. Και μετά βεβαίως αυτό αλλάζει τα πάντα ε, κύριε Τούρμες, έτσι δεν είναι το ίδιο το το 27 με το 30 πόσο φιλόδοξοι είμαστε παραδείγματο χάρη για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ξέρω ότι δεν θέλετε πάρα πολύ να το ανοίξουμε αν δηλαδή θα πάει στην οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας ή στην οδηγία περί κτηρίων, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, και τις οδηγίες που ισχύουν τώρα για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Αν δείτε το τι κάνω κάθε μήνα. Ε, κάθε μήνα ξεκινάω διαδικασίες επί παραβάση. Και δεν είναι και πολύ ευχάριστο για έναν επίτροπο γιατί μετά προσπαθώ να είμαι σε επαφή με τα μέλη και από την άλλη κινούμε διαδικασίες ε, για παραβασία. Αλλά οι οδηγίες αυτές λοιπόν που έχουν τα περισσότερα προβλήματα στην εφαρμογή είναι οι οδηγίες αυτές για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τα κτίρια. Λοιπόν, για τις τιμές του πετρελαίου Είναι πολύ πιο δύσκολο βέβαια να αναπτύξουμε ανανεώσιμε φύγε όταν είναι τόσο χαμηλή τιμή ή το πετρελαίο. Γιατί μετά θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να... Έχουμε μία δέσμευση για να επιτύχουμε τους στόχους του COP21 και δυσκολεύουν τα πράγματα με χαμηλές τιμές. Πόσο θα κρατήσει αυτό, ποια θα είναι η ικανότητα του Ιράν να έρθει στην αγορά, πώς θα ισορροπήσει η αγορά στο μέλλον υπάρχει συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ρωσίας και Ιράν θα συνεχίσει το μέλλον. Δύσκολο να πει κανείς. Αλλά εμείς πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως ε, των τιμών του πετρελαίου γιατί αν να περιμένουμε τις τιμές του πετρελαίου χαθήκαμε. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε, να δούμε το τι θα κάνουμε με τα βιοκαύσιμα στο μέλλον και ποιο ποσοστό θα πρέπει να ορίσουμε για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας. Για το LNG στην Μεσόγειο είχαμε κάποιες ερωτήσεις. Για την Gazprom θα, θα απαντήσω στο τέλος. Γιατί πιέζει ο χρόνος, θα πω λίγα λόγια όμως. Yeah, ε, δεν ξέρω αν προτιμάτε, να απαντήσω τώρα. Για την Κάσπρομ έχω μια ξεκάθαρη γραμμή που την είχαμε πάντα. Και είναι σαφής. Ε, Οποιοδήποτε αγωγός φυσικού αερίου πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάχνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ενέργεια, το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες. Και η Κομισιόν θα διασφαλίσει την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Είναι γεγονός πως λάβαμε την πρώτη αξιολόγηση για το εάν μπορεί να εφαρμοστεί το τρίτο πακέτο από την ε, νομική υπηρεσία της Κομισιόν και έχουν τεθεί σημαντικά ζητήματα τα οποία συζητάμε εσωτερικά και όταν έχουμε μια σαφή εικόνα θα έρθω στην Επιτροπή σας να σας πω ποια είναι η θέση μας. Να πω όμως το εξής. Οι νομικές πτυχές δεν είναι το παν γιατί οι πολιτικές και οι οικονομικές στοιχείες όπως ο αντίκτυπος της αγοράς, οι συνέπειες ε, της διαφοροποίησης ε, της ε, ασφάλειας της παροχής, επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί αν γίνει αυτός ο αγωγός, 80% του ρωσικού αερίου θα πάει σε έναν αγωγό. Ε, αυτό είναι κάτι το σημαντικό, αλλά βεβαίως, οπωσδήποτε, ε, η γερμανική αγορά θα περάσει από 40% σε 60% ρωσικό αέριο και θα έχουν πολύ πιο κυριαρχή θέση. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Αν η Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι χώρα διαμετακόμισης, όλες αυτές οι παράμετροι μαζί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η Κομισιόν για να διαμορφώσουν την κατάσταση. Όπως σας είπα, η Ουκρανία, ο σεβασμός του κοινοτικού δικαίου και βεβαίως ε, και η τιμή στην κάθε χώρα επιβαρύνεται και με τέλη διαμετακόμισης. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε τις συμβάσεις. Ε, δεν θέλουμε να μπλέκουμε εκεί που δεν μας παίρνουν, αλλά να πρέπει να ξέρουμε τους κινδύνους. Γι' αυτό έχουμε και το στόχο του 40%. Δηλαδή, για να ξέρουμε αν ε, υπάρχει κάποια επίδραση σε μια αγορά. Μετά ε, ετέθη το ζήτημα των περιφερειών. Να σας πω κάτι το είναι σημαντικό. Οι περιφέρειες και μετά θα περάσει τη Μάλτα και την Κύπρο. Οι περιφέρειες ε, που έφτιαξε η Κομισιόν έγιναν με βάση αντικειμενικές παραμέτρους αλλά δεν είναι κάτι το θέσφατο, είναι κάτι το οποίο συζητάμε με το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη. Κάναμε μια αρχική χάραξη των περιφερειών και αν δείτε στα παραρτήματα το τι έχουμε κάνει, στα βορειοδυτικά υπάρχει η Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, μετά Μπενελούξ, Ολλανδία, Γαλλία, Βουλγαρία, μετά το νότιο διάδρομο Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, μετά Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, μετά Αυστρογκαρία, Σλοβενία, Ιταλία, Βαλτική και Φιλανδία και μετά Δανία, Σουηδία. Η Κύπρος από μόνη της δεν διασυνδέεται με τίποτα και η Μάλτα το ίδιο αν διασυνδεθεί η Μάλτα με άλλο κράτος μέλος ε, θα πάει σε άλλη περιφέρεια. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό. Ε, δεν μπορεί. Εντάξει, αν θέλει μια χώρα να πει δεν θέλω να είμαι σε αυτή την περιφέρεια, να είμαι στη δίπλανη, ναι, εντάξει, θα είναι μια πολιτική απόφαση. Εμείς κάναμε μια πρώτη πρόταση. Με βάση τις υφιστάμενε περιφερειακέ αγορές, ε, το βαθμό διασύνδεσης, τη γεωγραφία προφανώ Αυτέ οι παραμέτρους. Οπωσδήποτε τώρα για την Κύπρο και τη Μάλτα θα πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε την απομόνωση, να, υπάρχουν, να υπάρχει πρόσβαση σε τρεις πηγές αερίου και πρέπει να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη ε, και τα νέα ευρήματα στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα έχουν τα σχέδια των αγωγών. Να απαντήσω στην κυρία Κάπελ που είπε πώς θα συνδυάσουμε την ευελιξία. Υπάρχει λοιπόν ε, σε κάποιες αγορές σύνθημα ευελιξίας ε, και η σχέση με τις αγορές ηλεκτρισμού. και δεν έχουν και κάποιο επαρκέ επίπεδο φιλοδοξίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υπάρχει και μια αποκεντρωμένη παραγωγή. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί κάποια ευελιξία σε αυτή την αγορά. Και εκεί πέρα θα χρειαστεί πράγματι κάποιο μέσο ανάγκης και πιθανότητα αυτή η πηγή παραγωγής θα είναι το φυσικό αέριο. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα με τις ε, στενοπούς στον τομέα του φυσικού αερίου. Δεν μιλάμε για κατασκευή μεγάλων αγωγών. Όταν η Ρωσία πήρε την απόφαση να ακυρώσει τον South Stream και μας ε, το είπε, μας είπε το 2019 θα φέρω φυσικό αέριο στα σύνορα της Τουρκίας και η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει άλλο αγωγό, είπαμε όχι, θα κάνουμε διασυνδέσεις και αντίστροφες ροές. Γι' αυτό, αν δείτε, εργαζόμαστε κυρίως σε τρεις ομάδες. Σε κεντρική και νότια Ευρώπη υπάρχουν έξι έργα προτεραιότητας με δύο βασικούς διαδρόμους από Ελλάδα προς Βορρά και έναν οριζόντιο. Στην Βαλτική επίσης έχουμε έξι έργα προτεραιότητας για αποθήκευση και διασύνδεση των τριών Βαλτικών με τη Φιλανδία και Νοτιοδυτική Ευρώπη δύο έργα, ένα με την Πορτογαλία και ένα που διασχίζει τα Πυρηναία. Οπότε προσπαθούμε, όπως είπα, να ξεπεράσουμε τις ε, στενοπούς, γιατί το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε περισσότερα εργοστάσια LNG, έχουμε ήδη αρκετά. Είναι εκεί πέρα που λείπουν οι διασυνδέσεις για να έχουμε έτσι ένα δίκτυο. Θα έχουμε λοιπόν μια ευέλικτη αγορά και θα έχουμε ως ρεζέρβα το φυσικό αέριο. Οπότε, κύριε Τούρμες, στο επίπεδο που θα χρειαζόμαστε όντως στο μέλλον, Εάν έχουμε φιλόδοξες πολιτικές ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας οπωσδήποτε θα χρειαστούμε λιγότερο ψικό αέριο. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε το επίπεδο φιλοδοξίας και μπορεί το Κοινοβούλιο να είναι πιο φιλόδοξο από εμάς. Αλλά και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι φιλόδοξος. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Um, Έχω τώρα ένα κατάλογο μιλητών. Μπενίντο Είναι ο πρώτος. Δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, ε, είπατε ότι έχουμε τη συμφωνία COP21. Ε, αποφάσισε αυτή η συμφωνία να μειώσει δραστικά τα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το LNG. Αλλά αυτό έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με αυτούς τους στόχους. Είναι εναλλακτική πηγή ε, ενέργειας. Λέτε θα μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα αξιολογήσουμε όμως αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να δούμε α, τη διαδικασία α, σε όλες τους τις ε, φάσεις από την εξόριξη, τη διήλυση, την υγροποίηση, τη μεταφορά, την καύση για να καλυφθούν και στρατηγικοί στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, το να αλλάξουμε δηλαδή τις ε, ε, συμμαχίες και την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκεκριμένες χώρες. Όμως δεν γλιτώνουμε από τις πολύ σοβαρές ε, περιβαλλοντικές ε, συνέπειες. Θα πρέπει να επενδύουμε στην ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία. Δεν θα πρέπει οι στρατηγικοί αυτοί οι λόγοι να υπερισχύσουν. Να μην στηρίξετε το φυσικό αέριο όπως στηρίξατε τις εξορρυκτικές βιομηχανίες, τις βιομηχανίες εξόρυξης πετρελαίου και ουρανίου μέχρι τώρα κύριε Κανιέτε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, παρουσίαση του με την οποία ξεκαθάρισε κάποια θέματα ε, τα οποία είχα κάποιε απορίε ε, για να εγγυηθούμε ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου και προσιτέ για όλου του καταναλωτέ. Πώ θα πετύχουμε αυτό το στόχο, εάν δεν υπάρχει φυσική ενοποίηση και ολοκλήρωση των αγορών. Έχουμε το φυσικό, το ευρωπημένο αέριο, ε, τη δυναμικότητα των μονάδων στην Ευρώπη. Αρκούν για να καλύψουν την, την ευρωπαϊκή ζήτηση. Δεν έχουμε ω πρόκληση να δημιουργήσουμε μια συστοιχία νέων μονάδων, αλλά πρώτα απ' όλα να στοπίσουμε τις υφιστάμενες μονάδες και να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις. Μας το είπε και ο Επίτροπος. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω την περίπτωση της Ιβερικής Χερσονήσου. Είναι ένα παράδειγμα, έχουμε οκτώ ε, μονάδες ε, υγροποίησης και μπορούμε να μειώσουμε έτσι την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της Ιβερικής Χερσονήσου. Το να προχωρήσουμε το μικάτα μέσω της Καταλωνίας θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε 14 ε, δις ε, κυβικά μέτρα ε, ως δυναμικότητα. Άρα πολύ μεγαλύτερη η συνεισφορά από την Ισπανία για την ορφαδιασμό της Ευρώπης. Επίσης, το κόστος της μηνοποίησης αγοράς που θα το φέρει οι καταναλωτές της Ιβυρική Χερσονήσου ανέχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα το κόστος της μη ενοποίηση και η έλλειψη σύγκληση των τιμών και στην Ιβυρική Χερσονήσου αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές είναι νομίζω λόγος ικανός και επαρκής που θα δικαιολογούσε τις μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενοποίηση των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ε, κυρία Μπέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Λίγες σύντομες παρατηρήσεις από μένα. Μιλάτε για περιφερειακή συνεργασία και αυτή την πρόταση ακολουθεί, αυτή τη λογική ακολουθεί και η πρότασή σας. Θετικό αυτό, γιατί έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε περίπτωση ανάγκης. Όμως, είπατε πως είναι μόλις μία πρώτη πρόταση αυτή και εγώ δεν συμφωνώ με την πολύ αυστηρή χάραξη των περιφερειών. Π.χ. λέτε πως ε, η Γερμανία πάει μαζί με Τσεχία, Σλοβακία και Σλοβακία. Μα έχουμε πολλές γειτονικές χώρες. Δεν θα γίνει καμία πρόβλεψη εκεί πέρα. Μετά, μιλάτε για τους προστατευμένους ε, πελάτες και λέτε πως χρειάζεται ξεκάθαρος ορισμός ποιοι είναι οι προστατευμένοι πελάτες. Το ίδιο χρειάζεται για όλους νομίζω. Μετά για τις συμβάσεις ε, κρατών ε, μελών με επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Έχουμε εδώ πέρα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που μας δίνει κάποια εργαλεία και η Κομισιόν θέλει να ε, βλέπει τις συμβάσεις που είναι τουλάχιστον ενός έτους και 40% και λέτε πως Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε η Κομισιόν στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται να ζητήσει από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν και άλλες συμβάσεις. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αν θέλει η Κομισιόν να βλέπει ιδιωτικές συμβάσεις θα πρέπει να έχει πολύ καλή αιτιολόγηση. Επίσης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που ελπίζεται από μια τέτοια διαφάνεια. Πράγματι, κάποιες χώρες είναι εξαρτημένες 100% από συγκεκριμένους ορμηθευτές Το να δείτε τη σύμβαση όμως δεν το αλλάζει αυτό. Η διαφάνεια δεν ξέρω αν είναι γεωπολιτικό εργαλείο και στέλνει μήνυμα προς την Ρωσία. Ε, εμένα θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω για το αν αυτό θα οδηγήσει όντως σε καλύτερους όρους ε, της σύμβασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πολύ. για την παρουσίασή σας, κύριε Επίτροπε. Και σας συγχαίρω για τις προτάσεις σας που νομίζω ότι συνιστούν και θα αποτελέσουν σημαντική πρόοδο. Εάν θέλουμε να έχουμε ανεφοδιασμό από διαφορετικές πηγές, αυτά τα μέτρα θα πράνε προτεραιότητά μας. Και για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού ε, το να έχουμε περισσότερες από μία πηγές, αυτό είναι σημαντικό. Ε, ακούσαμε από την Κομισιόν ε, ότι χρειάζεται συμπληρωματικότητα στο σχεδιασμό της αγοράς και θα πρέπει να εστιάσουμε στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει οι ορυκτές, τα ορυκτά καύσιμα να είναι όλο και μικρότερο το ποσοστό του στο ενεργειακό μείγμα. Εάν θέλουμε να περάσουμε σε μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα θέσω ένα προφανές ερώτημα, αλλά ε, σημαντικά, σημαντικό ερώτημα για το πολιτικό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικοί προμηθευτές ε, φυσικού αερίου στα σύνορα της ε, Ευρώπης. Μην, ξεχνάσουμε όμως, μην ξεχνάμε όμως και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για ανεφοδιασμό και για συμπληρωματικότητα στα δυτικά και μπορεί να εξασφαλίσουν και μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά και μεγαλύτερη διαφάνεια. Όπως είπε και ο συναδελφό μου, ε, η Δυτική Χερσόνησο είναι μία από τις παραγωγούς περιοχές. Έχει θαυμάσια πρόσβαση διαθαλάσση, όχι μόνο μέσω Μεσογείου αλλά και μέσω Ατλαντικού και μπορούμε δυνητικά να διευρύνουμε την εμβέλειά μας και έτσι μπορούμε να ε, δώσουμε φυσικό αέριο ούτω ώστε να υλοποιήσουμε την παγκόσμια στρατηγική μα για το φυσικό αέριο. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίε και εσείς βέβαια είστε ευρωπαϊκό επίτροπο, αλλά, γιατί εδώ μιλάμε για μια χώρα ουσιαστικά. Αλλά τι γνώμη έχετε για την αγορά της Ιδρυκή Χερσονήσου, ε, τι μέλλον έχει. Ευχαριστώ. Η Μούντι. Thank you very much. And, uh, yeah. Ευχαριστώ. Στοιχεία του πακέτου είναι πάρα πολύ θετικά, βέβαια. Θα ήθελα να θέσω όμως ένα συγκεκριμένο σημείο. Πρώτη, το πρώτο πακέτο δράσης ε, μετά το Παρίσι εστιάζει σαφώς στο φυσικό αέριο. Ενώ, όπως είπατε, η δράση για τη μετάβαση σε μια νέα ενεργειακή αγορά χρειάζεται χρόνο. Και άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατόν, να δρούμε το συντομότερο δυνατόν. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό που ακούστηκε. Ότι τώρα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε αυτή τη μετάβαση σε αυτή τη φάση τώρα. Το θέμα της ε, περιφερειακής συνεργασίας είναι το δεύτερο. Και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία αυτή. Μιλάμε για αυτήν, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να την υλοποιήσουμε. Τέλος. Μιλήσατε για το ΕΦΣΙ επίσης και το ΣΥΕΦ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πώς θα υποστηρίξουμε τις περιφερειακές πλατφόρμες μέσα στα κράτη-μέλη παρά τις ε, υπερεθνικές περιφερειακές ε, πλατφόρμες και δυνατότητα να δούμε εναλλακτικέ εναλλακτικά μοντέλα. Ενέργεια παράγεται συνεταιριστικά, ας πούμε, σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και διάφορα προγράμματα και έργα ε, εξασφάλισης ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο κύριος Ταζανόφσκι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έχουν ε, απαντηθεί. Μία θέλω να θέσω μόνο. Αναφέρατε τη σημασία των ε, εργοστασίων που χρησιμοποιούν ε, φυσικό αέριο. Ε, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και για να σταθεροποιήσουν το σύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά στην πραγματικότητα τέτοιου τύπου εργοστάσια δεν έχουν χτιστεί. Δεν ξέρω πολλά τέτοια εργοστάσια. Καταρχάς, ε, η τιμή του αργού πετρελαίου και γενικά τις ε, ενέργειες που χρησιμοποιείται αρχικά για αυτά. Επίσης, επειδή δεν θα ξέρουμε πόσο συχνά θα χρησιμοποιούνται η ενέργεια που, παρουσιάζεται από αυτά, που παράγεται από αυτά τα εργοστάσια. Ε, το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό για, στο Κοινοβούλιο και είμαστε πάντα στο ίδιο, στην ίδια κατάσταση. Και η κατάσταση είναι εξή, ότι τη σταθερότητα στο δίκτυο την εξασφαλίζουν τα εργοστάσια τα οποία ε, χρησιμοποιούν α, άνθρακα και όχι φυσικό αέριο. Δεν θα πρέπει να αναδιαμορφώσουμε τις στρατηγικές μας σε ό,τι αφορά ε, και τα τέλη που επιβάλλουμε για να σταθεροποιήσουμε το δίκτυο. Η κυρία Σπυράκη. Thank you, Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Κανιέτε. Θα ήθελα να επιμείνω στο συμπέρασμά σα ότι οι ειδικέ συμφωνίε ε, υπογράφηκαν, ε, που υπογράφηκαν στο παρελθόν δεν είναι ικανοποιητικέ. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια μετατόπιση από το κράτο μέλο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τις διαδικασίες επί για την οποία αφαιρθήκατε. Ποια είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά τις ευιστάμενες συμφωνίες μεταξύ κρατών μέλων και διακυβερνητικών. Αν θέλει παράταση της Ευρωπαϊκής συμφωνίας ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Κομισιόν και αν όχι, η στρατηγική της Κομισιόν πώς θα επιτευχθεί. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα για τις καλύτερες διασυνδέσεις. Είπατε ότι θα εστιάσετε στις πραγματικά σημαντικές διασυνδέσεις. Αυτό επιτόπου πώς θα το πετύχετε. Θα ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τα επιχειρησιακά του σχέδια στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για να ξεκινήσουν την ανάπτυξη ίσως αγωγών ή αποθήκευσης ε, καλαμικών συνόρων. Ευχαριστώ. Thank you very much, σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Δεν βλέπω κάποιον. Α, κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την αρχή της ε, ε, διασύνδεσης και αναφερθήκατε σε κάποια κράτη-μέλη. Μιλήσατε επίσης ε, για τη σχέση κόστους ωφέλους. Έχουμε το θέμα των πηγών ενέργεια, έχουμε το θέμα των προσιτών τιμών. Εκεί όμω τι γίνεται με τη σχέση κόστου-οφέλου, θα γίνει προβληματική η σχέση αυτή. Μήπω λοιπόν η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα τη σχέση κόστος-οφέλους. Μιλά για τις διασυνδέσεις πάντα. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε μια πολιτική απόφαση που θα τη στηρίζει η Κομισιόν. Just a follow-up question. Κύριο Στούρμέ, ε, να δευτερολογήσω και να κάνω μια ακόμη ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για στατική LNG λέγοντα ότι ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΦΣΙ και του ΣΕΦ. Να σας υπενθυμίσω ότι στην νομοθεσία περί ΣΕΦ λέγεται ότι μόνο το 5% μπορεί να πάει στο φυσικό αέριο. Γιατί όταν διαπραγματευτήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη αυτή την ε, συμφωνία για το Connecting Europe, αυτό που θέλαμε ήταν να δοθεί προτεραιότητα στις υποδομές ηλεκτρισμού. Γνωρίζουμε από πέρυσι ότι έχουν ε, χρηματοδοθεί κάποια project για το φυσικό αέριο. Εμείς όμως πρέπει, και ελπίζω να μην το λέω μόνο για τον εαυτό μου, πρέπει να τηρούμε κάποιες δεσμεύσεις. Στην νομοθεσία προβλέπεται 50%, όχι παραπάνω για το φυσικό αέριο. Πώς μπορείτε να υπόσχεστε 50% εάν ήδη έχουν πάει εκεί τα περισσότερα κονδύλια και δεν μας έχουν μείνει πολλά κονδύλια για τον ηλεκτρισμό. No other request for floor. Δεν έχετε ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, κύριε Επίτροπε. Πολλά είναι τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Για τον κύριο Μπενίτο Θουλουά. Είναι σαφές ότι η COP21 η συμφωνία για να ανακοπεί η υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κατά τους δύο βαθμούς ε, Κελσίου 1,5 ε, βαθμό ουσιαστικά είναι ο στόχο, μα οδηγεί ε, στην πλήρη απαλλαγή τη οικονομία από τον άνθρακα μέσα σε αυτόν τον αιώνα. Και μία από τι δεσμεύσει όλων των μερών και φυσικά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 2020 να τεθεί επιτάπητο ε, στρατηγική για το, την αλλαγή του κλίματος και οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξες από τις αναπτυσσόμενες και θα έχουμε πολύ σημαντικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών. Πάρα πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντική στόχη. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το 2030 θα είναι πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο, είναι προφανέ ότι θα είναι λιγότερο και αρκετά λιγότερο σημαντικό το 2050. Είναι προφανέ αυτό, ε, είναι αυτονόητο. Όταν λοιπόν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε υποδομές Κύριε Τούρμης, δεν έχουμε στόχο να βάλουμε μεγάλα μακρόπνοα project επιτάπητος. Θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι διευθυντές που λείπουν και είναι απαραίτητες για να εγγυηθούν ε, τον επαρκή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα προχωρούμε αυτή τη διαδικασία απαλλαγή από τον άνθρακα. Να πω τι είπε ο κ. Μπλάκ και ο κ. Ζωρίνιο. Είναι προφανές ότι δεν έχει νόημα να έχουμε ήδη ε, αυτές τις ε, τεράστιες ε, και πάρα πολύ καλά διανεμημένες διάσπαρτες μονάδες υγροποίησης σε κάποια λιμάνια που είναι πολύ καλά, σε πολύ καλά σημεία από γεωγραφικής πλευράς, αλλά δεν μπορεί να τι αξιοποιήσει πλήρω η Ευρωπαϊκή Αγορά, γιατί δεν έχουμε τη διασύνδεση στα Πυρηνιά και επειδή ο οριζόντιο άξονα στη Γαλλία δεν έχει επικοινωνία με την Ανατολική Αγορά. Δεν χρειάζονται λοιπόν αυτέ οι μεγάλε υποδομέ. Θα δείτε ότι στον ηλεκτρισμό ουσιαστικά επενδύουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά υποδομέ για το φυσικό αέριο, αυτέ τι αναπτύσσει κυρίω ο ιδιωτικό και όχι ο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιο τομέα όμω έχει δύο στοιχεία παρέχει την χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΦΣΥ και κατά δεύτερον για να βγουν οι λογαριασμοί μπορεί να δίνει ε, κάποια χρηματοδότηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Διασύνδεση για να έχουμε αποδοτικά project. Εμείς κινούμαστε ε, με όρους σύνεσης, οφροσύνης. Δεν θέλουμε έκρηξη φυσικού αέριου. Το αντίθετο, ε, εμείς εγγυόμαστε ότι ναι να αναπτύσσουν περισσότερο τις ανανεώσιμε και αυτό είναι ο στόχος μας, έχουμε εφεδρικά αυτή την ε, ανάπτυξη του φυσικού αερίου. Ήδη πάνω από το 50% ε, θα θέλουμε να το παράσχουμε με τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θέλουμε και 80 και 90% να πετύχουμε, αλλά κάποιε ημέρε έχουμε μεγάλη ευμεταβλητότητα και διακύμαση. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ένα εφεδρικό μηχανισμό. Το θέμα είναι αυτού του μηχανισμού εφεδρικού πώ του χρηματοδοτούμε. Έχουμε τι ε, μονάδε συνδυασμένου κύκλου ή αυτέ τι μονάδε που παράγουν άνθρακα και ανάλογα χρησιμοποιούμε. Το ενεργειακό σύστημα δηλαδή, πώ εγγυάται ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά οι καταναλωτέ να έχουν στο σπίτι του ε, ενέργεια ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η Επίτροπο ε, Ανταγωνισμού κάνει μια πρόταση και θέλει να δει αν ε, ε, στηρίζουν τα κράτη-μέλη αυτέ τι ε, πληρωμέ αναδυναμικότητα, μήπως υπάρχει στρέβλωση ε, του ανταγωνισμού. Και θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα, να βρει έναν τύπο η επιτροπή η Αρμόδια για να δει πώ θα το ρυθμίσω αυτό το ζήτημα. Είναι προφανές όμως ότι όσο αναπτύσσουμε τι ανανεώσιμε και αναβάζουμε την ενεργειακή απόδοση, όλο θα μειώνονται οι ανάγκες ενέργειας και θα υπάρχουν πολλές μονάδες που θα παραμένουν ε, απαρχαιωμένες και θα πρέπει να ε, διαλυθούν, να κλείσουν. Και δεν μιλάμε για κάτι πολύ ε, άμεσο, μιλάμε με την προοπτική το 2050. Και φυσικά κάθε χώρα πρέπει να ε, καθορίσει το δικό της ενεργειακό μείγμα και την παραγωγή της ενέργειας. Η Κομισιόν από την πλευρά της πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις για όλες τις χώρες. Εγώ δεν λέω ότι είμαι υπέρ του πετρελαίου, κάποιος το υποστήριξε. Όχι, εγώ το μόνο που αναζητώ είναι να έχουμε στον πιο καθαρά ορυκτά καύσιμα, να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα μας επιτρέψουν ε, να χρησιμοποιούμε τα ορυκτά καύσιμα ως εφεδρική πηγή ενέργειας αν έχουμε ζήτημα με τις ανανεώσιμε. αν δεν έχουμε αρκετό ήλιο, ηλιοφάνεια, αν δεν φυσάει αρκετά κάποια μέρα. Ε, και αυτή νομίζω είναι η λογική τη COP21 Μα μου είπατε ότι τώρα μετά την ΚΟΠ ε, μας ε, προτείνεται μία δέσμη για το φυσικό αέριο. Πριν από την ΚΟΠ είχαμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιωμάτων Εκπομπών. Αυτό ήταν το πρώτο πακέτο που καταθέσαμε, το ETS πριν την ΚΟΠ και στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλαμε να βάλουμε μια τιμή στον άνθρακα. Σαφές. Το δεύτερο πακέτο Α, και αμέσως ήρθε αυτό, ήταν ανώσιμε πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και έχουμε και ένα άλλο, ένα πρόστο πακέτο που έρχεται, πολύ διαφορετικό από αυτό. Είχαμε όμως τα προβλήματά μας με την Ουκρανία. Μας είπαν κάποιε χώρε θα παρακάψουν την Ουκρανία. Μιλάμε μετά για τα τουρκικά σύνορα και το φυσικό αέριο. Ο κ. Πίτρο Εύκοβιτ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με τη ε, διαπραγμάτευση του χειμερινού πακέτου για να έχει Ουκρανία αέριο το χειμώνα. Ξέρουμε λοιπόν ε, ότι θέλουμε να έχουμε πολύ πιο αξιόπιστου και έχουμε την ε, Νορβηγία για παράδειγμα. Αλλά ε, κάποιοι άλλοι προμηθευτέ από καιρού καιρών μα δημιουργούν κάποιε αμφιβολίε και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ο κ. Μπλάνκο πολύ καλά τα είπε ότι δεν έχει κανένα νόημα πράγματι οι διασυνδέσεις μέσω των Πυρενέων, ανατολικό σε τρίτο άξονα μέσω τη Πορτογαλία, ε, να αναπτυχθούν αλλά να έχουμε ε, μια ε, Ιβερική χερσόνησο που δεν συνδέεται. Πρέπει να συνδέεται πλήρως με την υπερωτική Ευρώπη και ιδίω αν δείτε την καμπύλη των τιμών. Αν δείτε την καμπύλη των τιμών θα δείτε το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και από τους αγωγούς φυσικού ε, Οι τιμές πλησιάζουν πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ, επειδή ε, υπάρχει αναπροσαρμογή των τιμών φυσικού αερίου στην τιμή του περετρελαίου. Και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αντιστοιχεία στις τιμές και έχουμε κοιτάσματα ε, στο Μεσόγειο, στα Νότια Σύρο, πάρα πολύ σημαντικά, επομένως έχει κάθε νόημα. Για την κυρία Βέρνερ που μίλησε για την περιφερειακή προσέγγιση και ποια θα είναι η αντίδραση των κρατών μελών. Ακούστε, πρόκειται για φιλόδοξη πρόταση. Η Κομισιόν αυτό πρέπει όμω να διατυπώνει, φιλόδοξε προτάσει. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει το θέμα αυτό. Έχουμε διάλογο. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε όπω κάναμε στο παρελθόν. Ή θα εργαστούμε σε περιφερειακό επίπεδο, με αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι άλλη εναλλακτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί βασίζεται, στην αλληλεγγύη. Έχουμε την μεταναστευτική κρίση και το στοιχείο τη αλληλεγγύη. Ε, εδώ ίσως να μην είναι και στη μεγαλύτερη φόρμα. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού και του εφοδιασμού εν γέννη, χρειάζεται έλεγγυη. Αυτό είναι σαφές. Και γι' αυτό έχουμε τις ανάδρομες ροές και γι' αυτό εμείς προτείνουμε αυτή τη φιλόδοξη προσέγγιση. Και νομίζω ότι και κατά το παρελθόν έχουμε κάνει αυτές τις προτάσεις που κάνουμε. Και με τις διακυβερνητικές συμφωνίες τι έγινε. 124 είχαμε. Το 1 τρίτο ε, τι είπαν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γιατί ε, το τάδε κράτο δεν θέλει να στο τραπέζι να διαπραγματευτούν και καλά τα λέγανε. Πάμε στο δικαστήριο για το τίποτα. Τώρα έχουμε την εξάντε αυτή αξιολόγηση, οπότε μπορούμε να πω στο κράτο μέλο μην το κάνετε. Αυτό προσπαθήστε να αλλάξετε κάπως τα πράγματα γιατί έχετε χρόνο τώρα στη διάθεσή σας. Βέβαια, Εάν υπάρχει μια ε, ισχύουσα ε, διακυβερνητική και θέλουν να την αναδιαπραγματευτούν, πρέπει να τηρηθούν οι σημερινές ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των διακυβερνητικών συμφωνίων. Αν παρεμβαίνουμε πολύ ή όχι τελικά, αν αναμειγνιόμαστε. Ακούστε, για να κάνουμε μια πραγματική μελέτη αντικτύπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πρέπει να ξέρετε ότι Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια είναι τα μέγιστα ε, ημερήσια ποσά, πού ε, φτάνει το αέριο, ποιος είναι ο όγκος, ε, ποια είναι η δυναμικότητα και χωρητικότητα και των διαφόρων επιχειρήσεων. Επομένως, εμείς λέμε ότι δεν αναμειγνιόμαστε υπερβολικά, γιατί εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα, δεν θέλουμε να ξέρουμε την τιμή άλλες αρχές θα δουν το θέμα των τιμών. Αν δείτε τον κανονισμό, αυτό το οποίο ζητούμε είναι πολύ σαφές. Για να το βρω, για να το βρω. Τι λέει εδώ πέρα. Διάρκεια, όγκος, σημεία, ε, ελάχιστη ό, κτλ. κτλ. Κάποιες προϋποθέσεις για να Ναι, εντάξει. Αλλά μετά αν θέλουμε να κάνουμε μελέτη αντικτύπου σε ανακράτος μέλος ε, ή μια ολιστική μελέτη αντικτύπου, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι σημαντικές συμβάσεις και ποια είναι η δυνατότητα προμήθειας και φοδιασμού που υπάρχει. Αυτό κάνουμε. Δεν χώνουμε τη μύτη μας. Για την κυρία Μούντι που μίλησε Κοιτάξτε, για μετά το Παρίσι. Πρέπει να ανταλλάξουμε όλα μετά το Παρίσι πλέον. Μεταφορές γεωργία κτίρια είναι τα πιο δύσκολα. Εάν πιστεύατε ότι το ETS ήταν δύσκολο, πλανάστε πλάνη ικτρά. Ήδη έχω ξεκινήσει ε, τα ταξίδια μου με την Πολωνία ξεκίνησα και σας λέω ότι αυτά που σας είπα είναι ακόμα πιο δύσκολα ζητήματα και θα είναι πολύ μακροχρόνιες οι συζητήσεις διότι εδώ έχουμε στόχους για κάθε κράτος μέλος. Και κάθε κράτο μέλο πρέπει να επεξεργαστεί αυτού του πολύ δύσκολου τομεί. Όμω θα έρθουμε με μια οδηγία και για την ενεργειακή απόδοση και για τι ανανεώσιμε. Θα έχουμε οδηγία και θα έχουμε και για τα ελαφρά φωτιά και τα οχήματα προτάσει ε, για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πολύ σύντομα θα τα έχετε όλα αυτά. Διασυνδέσεις. Να σας πω τι γίνεται αρχικά στον αγορά ηλεκτρισμού. Δεν δίνει σήματα για επενδύσεις. Υπάρχουν υποεπενδύσεις στον τομέα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή η αγορά ε, κοινοφελής υπηρεσίες δεν επενδύουν τίποτα. Ούτε σε νέους σταθμούς, ούτε στο δίκτυο, ούτε πουθενά. Άρα θα πρέπει ε, να δώσουμε όθηση. Για την ηλεκτρική ενέργεια πάντα. Τώρα, για, τη φυσική, για το φυσικό αέριο, η αγορά εδώ πέρα ε, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, λειτουργεί πολύ καλύτερα. Έχουμε τη στρατηγική LNG, μπαίνει περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά και νομίζουμε ότι αυτό είναι θετικό. Όμω ε, τα περισσότερα project ε, γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα, από ιδιωτικέ επιχειρήσει. Έχουμε πολύ μικρή στήριξη, 5,8. 5,85 κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του ΣΕΦ και Γι' αυτό θα πρέπει αυτό το περιορισμένο ποσό που έχουμε στη μα να το χρησιμοποιήσουμε πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στι περισσότερε ερωτήσει. Σίγουρα εφιλόδοξο το πακέτο. Σας διαβεβαιώνω όμω ότι και στην Επιτροπή είχαμε πολύ ε, μακρά συζήτηση. Επιλέξαμε αυτή τη φιλόδοξη προσέγγιση για το σχέδιο, τον ανασχεδιασμό της αγοράς. Ακριβώς το ίδιο. Θέλουμε πάλι να έχουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε, Επίτροπε. Χάρη στις δραστηριότητε σας μπορούμε και εμείς στην ε, Επιτροπή Ιτρέ να σκουμποθούμε, να δραστηριοποιηθούμε, γιατί έχουμε διάφορα θέματα να επιλύσουμε. Διάφορα πράγματα να πιέσουμε. Σας ευχαριστούμε να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε και σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τις πρωτοβουλίες σας. Όλες τις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστούμε και για τις πρωτοβουλίες για το κλιματικό πακέτο. Χαιρόμαστε που έρχονται τόσο συχνά στην Επιτροπή μας. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You will help me with Poland. <laughs> Uh, thank you, colleagues. Uh, last point for... Τελευταίο σημείο για σήμερα, συνάδελφοι. Μια μελέτη για την ανοιχτή καινοτομία ε, που συμπεριλαμβάνει και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Παρουσίαση από την Κριστίν Χάμζα και τον Τίτερ Ρέχφελτ από το ΜΕΤΙΣ. κατόπιν αιτήματο τη Επιτροπής Ήτρε έγινε αυτή η μελέτη. Αυτό να το τονίσουμε. Παρακαλώ σταματήστε τα πηγαδάκια, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. And uh, let me add, the study described... Να προσθέσω, η μελέτη αυτή προσθε... περιγράφει το πώς ε, μπορεί η ανοιχτή καινοτομία και η αποκεντρωμένη παραγωγή να ενισχύσουν την οικονομία μας. Και κάποιες συστάσεις, ναι, ναι. Στα διαφορετικά επίπεδα πολιτικής επίσης. Πώς δηλαδή θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ah, κυρία Χάμζα και ο κύριος Ρέφελτ. Λοιπόν, παρακαλώ να κάνετε την παρουσίασή σας. Έχετε 10 λεπτά. Μπορείτε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια πράγματα σε 10 λεπτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ανοιχτή καινοτομία και μελετήσαμε την ανοιχτή καινοτομία και την αποκεντρωμένη παραγωγή ταυτόχρονα. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές συνδέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρούμε πως υπάρχουν κάποιες παράλληλες εξελίξεις. Βλέπουμε πως ε, συνεισφέρουν στην ανανέωση της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, κυρίως στον τομέα της ε, παραγωγής, αλλά βεβαίως και όσον αφορά τον τομέα της υγείας, τον δημιουργικό κλάδο κτλ. Επηρεάζουν λοιπόν την διαδικασία με την ενσωμάτωση κοινωνικών πτυχών και ενδιαφέρον θα ήταν λοιπόν τα συνδυάσουμε αυτά την τεχνολογική πτυχή με την ε, κοινωνική πτυχή έχουμε λοιπόν ε, ένα συνολικό πλαίσιο και βεβαίως εφαρμόζονται σταδιακά αλλά υπάρχει η δυνατότητα να διαταράξουν τα υφιστάμενα πρότυπα υπάρχει Ε, λοιπόν, ένα όραμα το οποίο εξαρτάται από την ε, τεχνολογία. Λοιπόν, βλέπουμε σήμερα πως υπάρχει μια εφαρμογή σταδιακή η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπές μακροπρόθεσμα αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το αριθμιστικό περιβάλλον, τα επιχειρηματικά μοντέλα ίσως σε 30 χρόνια να κάνουμε μια αναδρομή και να πούμε πως εκείνη τη στιγμή έγινε η ανατροπή αλλά τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε Σύντομα η ανοιχτή καινοτομία απογειώθηκε στις αρχές ε, της δεκαετίας του 2000 ε, με βάση το έργο του Ασπάροφ αλλά βεβαίως ε, είχε ξεκινήσει η βιομηχανία τη δεκαετία του 1990 ορίζεται ως η επιταχυμένη χρήση εισρωών και εκροών για να υπάρξει μια αυξημένη χρήση της καινοτομίας στην αγορά. Βλέπετε πως δεν μιλάμε για καινοτομία μόνο από την πλευρά των χριστών αλλά και για κοινέ ε, επιχειρηματικές προσπάθειες, spin-in και spin-off. Δεν πρέπει λοιπόν να το μπερδεύουμε με την δωρεάν καινοτομία. Η ανοιχτή καινοτομία δεν είναι δωρεάν, είναι στην ιδιοκτησία των εταιριών και διαφέρει βεβαίως από την καινοτομία των χρηστών γιατί παραδείγματο χάρη τα ερευνητικά Ινστιτούτα, οι εταιρείε μπλέκονται σε πάρα πολλές βιομηχανικέ δραστηριότητες. Μέχρι στιγμή λοιπόν μιλάμε για τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και τώρα βεβαίως διαδίδεται και στις εταιρείες μέσης και χαμηλής ε, τεχνολογίας και ίσως εκεί πέρα θα διαδοθεί ευκολότερα γιατί δεν έχουν ξεχωριστά τμήματα τεχνολογίας και ανάπτυξης και έχουν μάθει να συνεργάζονται με τους ε, πελάτες τους. Η ανοιχτή καινοτομία λοιπόν είναι κάτι το πολύ ποικιλόμορφο, οι εταιρείε το βλέπουν με διάφορους ε, τρόπους και βεβαίως εξαρτάται αυτό από το επιχειρηματικό μοντέλο και υπάρχει ένα επίπεδο παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό. Θα επανέλθω σε αυτό. Πάμε τώρα στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Οι ρίζες τη τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκονται στη για του 1980. Τότε το έλεγαν γρήγορο, γρήγορα πρωτότυπα, μετά το έλεγαν προσθετική παραγωγή και βεβαίως τώρα μιλάμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση που γίνεται είτε σε ατομικό μεμονωμένο επίπεδο είτε κάπως πιο μαζικά. Η διαδικασία λοιπόν αυτή εκτύπωσης αναστρώμα ε, είναι η λεγόμενη τρισδιάστατη εκτύπωση και επειδή πρόκειται για μια προσθετική προσέγγιση εξοικονομούμε πάρα πολλά υλικά, ενέργεια κτλ. Μέχρι στιγμής ε, έχει εδρεωθεί και εδρεώνεται αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το καθημερινό πλέον, ειδικά στον τομέα των οδοντιατρικό, της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και υποτίθεται πως έχει την δυνατότητα να μας οδηγήσει σε κάποιες νέες βιομηχανίες και μακροπρόθεσμα αναμένουμε να μας οδηγήσει σε μια μετάβαση από τη μαζική παραγωγή σε μια μαζική και εξατομικευμένη παραγωγή. Η αλυσίδα της ε, αξίας, της δημιουργίας αξίας είναι πολύ αποκεντρωμένοι. Έχουμε τρεις ε, ομάδες. Έχουμε τους προμηθευτές των συστημάτων, ε, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, αυτά τα οποία αναφέραμε, αεροδιαστημική, οδοντιατρική κτλ. Και βεβαίω έχουμε την ε, κοινότητα του open source που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια. Το πρόβλημα είναι πως ε, η εφαρμογή της ε, τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ε, καινοτομίας στην παραδοσιακή βιομηχανία διαφέρει πολύ από την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Είναι θα έλεγα διαφορετικές κουλτούρες και είτε έχουμε είτε σύγκρουση είτε συνεργασία. Εδώ πέρα λοιπόν προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα διάφορα πλαίσια η ανοιχτή λοιπόν καινοτομία είναι μέρος του πώς θα επανεξετάσουμε και θα ξαναδούμε τις στρατηγικές μας για την καινοτομία, κοινωνική καινοτομία, το τι σημαίνουν όλα αυτά τα μοντέλα. Η βιομηχανική τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ενσωματωμένη στην βιομηχανία 4.0 όπως λέμε Πρόκειται λοιπόν για μία μόνο από τις ε, διάφορες ε, τεχνολογίες που υπάρχουν, τεχνολογίες ψηφιοποίησης. Η εκτύπωση τρισδιάστατη στο περιφερειακό επίπεδο είναι στο λεγόμενο κίνημα των Fablet. Και πάλι λοιπόν Μιλάμε και για άλλες τεχνολογίες όπως η κοπή με λέιζερ και τα λοιπά. Και βεβαίως ε, η ανοιχτή καινοτομία αφορά και το εάν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν κάποια περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας. Η κοινότητα open source ε, έχει ε, εμπλακεί και στα δύο και στο κίνημα των παραγωγών που βασίζεται στους ιδιώτες χρήστες. Μιλάμε δηλαδή για έναν εκδημοκρατισμό του καπιταλισμού, έχει τις ρίζες του στην Καλιφόρνια. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η έκφραση, αλλά μιλάμε για την διάδοση των τεχνολογιών. Στο μέσο βλέπετε τις διασυνδέσεις μεταξύ ανοιχτής καινοτομίας και ε, τρεις διάστατες εκτύπωσης μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες, οριακές ε, και βεβαίως μιλάμε στο θέμα των νέων αστικών βιομηχανιών και υπάρχει στενή σύνδεση στο βασικό επίπεδο όπως είπα μεταξύ των δύο. Λοιπόν, κάποιες προκλήσεις και συστάσεις. Το βασικό ζήτημα είναι το νομοθετικό και αριθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές ε, δραστηριότητες στο παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία είναι πως χρειάζεται μια ισορροπία. Αυτό εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου, του ρυθμιστικού πλαισίου για να δώσουμε κίνητρα και από την άλλη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα κάνει πιο εύκολες τις ροές της γνώσης. Το βασικό ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι το ζήτημα της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ε, και διάφορα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το να γίνουν πιο εύκολα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά από την άλλη και η ανοιχτή καινοτομία Βεβαίω το κίνημα, το open source, λέει πως η πνευματική διοκτησία έχει ξεπεραστεί και χρειάζεται ελεύθερη ροή της ε, γνώσης ε, μετά. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για νέες ε, επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις μέχρι στιγμής οι οποίες επιταχύνουν τις στρατηγικές ανοιχτής καινοτομίας. Κάποια από αυτά τα εργαστήρια, στην, ειδικά στην Ιταλία, ξεκινούν χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς επιχειρηματικά μοντέλα. Και βεβαίω υπάρχουν και συνέπειε στη λιανική, στον λιανικό τομέα, νέες δουλειέ κτλ. Και βεβαίω η εκπαίδευση και τα προσόντα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βασικό λοιπόν θέμα είναι πώ θα γεφυρώσουμε τι παραδοσιακή γνώση, τη μαστοριά που υπάρχει μαζί με την δυνατότητα για τεχνολογική εκπαίδευση. Συχνά βλέπουμε πανεπιστημιακούς και νέους να εργάζονται στο διαδίκτυο, να προγραμματίζουν, αλλά μακροπρόθεσμα το ερώτημα είναι πώς μπορούν να επανέλθουν στην παραδοσιακή κατεργασία των υλικών. Και βεβαίως οι περιβαλλοντικές πτυχές κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά το μιλάμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Δεν υπάρχει κάποια εικόνα για τον γενικό κύκλο ζωής και βέβαια υπάρχουν και οι περιφερειακές πτυχές, όπως είπα, για να δούμε τα περιφερειακά συστήματα καινοτομία που εστιάζουν παραδείγματος χάρη στις αστικές βιομηχανίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ρενφέλτ. Would like to, to give you one, question to, uh, mm-hmm. ask. Μία ερώτηση να σας κάνω για να τα απαντήσετε αμέσω. Συχνά λέμε ότι γεννηθήκαμε πριν από την νέα βιομηχανική επανάσταση και τη συνδέουμε ε, συχνά με τη ρομποτική. αυτή η ανοιχτή καινοτομία και η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι η βιομηχανική επανάσταση Παριθμό 5. Όχι. Η ρομποτική, το 3D printing είναι στοιχεία στη διαδικασία ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Δεν είναι το νούμερο 5, το νούμερο 6. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. γιατί πρέπει να έχουμε και μία σειρά σωστή με όλες τις ε, επαναστάσεις που λαμβάνουν χώρα. Κύριος Ταμπουράνο, σας ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη, τη διαβάσαμε πολύ προσεκτικά. Μάλιστα τη μεταφράσαμε και στα Ιταλικά, εγώ και το προσωπικό μου, ε, για να το στείλουμε στην Ιταλία, γιατί μόλις τώρα ε, γεννιέται αυτή η τεχνική, το 3D printing και γεννάει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους πολίτες. Όμω, έχουμε κάποιες ανησυχίες και κάποια ερωτικά, ερωτηματικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε διάφορους τομεί που αφορούν το θέμα αυτό. Καταρχάς μια επιστοποίηση των ε, συσκευών που μπαίνουν στα σπίτια μας. Έχουμε δηλαδή μικρά, ε, μικρά εργοστάσια ας πούμε μέσα στο σπίτι και δεν ξέρουμε τι εκπομπές παράγουν. Ε, και δεν έχουμε και στοιχεία για την ασφάλεια. Υπάρχει ας πούμε ε, ένας εκτυπωτής που αρχίζει να τίθεται στο εμπόριο για τα παιδιά στην Ιταλία. Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά γιατί δεν ξέρουμε διάφορα στοιχεία. Αυτά για τις συσκευέ. Αλλά δεν υπάρχει και επιστοποίηση ε, καθώς και επισήμαση ε, πάνω στα υλικά δεν ξέρουμε τι είναι, τα, τα, ας πούμε, τι είναι οι χρωστικές, ποια είναι τα έκδοχα ας πούμε, ε, διαφόρων ουσιών. Ακόμα και στον ιατρικό τομέα. Εγώ πριν έρθω εδώ ήμουνα ε, οδοντίατρος και υπήρχαν τεράστιε τεράστιες και στα, στα προσθετικά αλλά και όλο το υλικό που χρησιμοποιεί ένας οδοντίατρος ε, έχει αλλάξει, αλλά δεν υπάρχει πιστοποίηση ε, για το υλικό που χρησιμοποιεί ο δοντίατρο και που βάζει το ανθρώπινο σώμα. Έπειτα, ο κύκλο ζωή. Πώ παράγονται αυτά τα υλικά, ποια είναι η διαδικασία, η αλυσίδα και τι δυνατότητε έχουμε ε, στα πλαίσια τη ε, κυκλική οικονομία, δηλαδή ανάκτηση του πλαστικού, ούτω ώστε να παράγουμε τα, τα νέα υλικά με την σειρά του. Μπορείτε να μα πείτε κάτι παραπάνω, εσεί πάνω σε όλα αυτά. Και αν στο μέλλον έχετε περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας να τις ε, λάβουμε για να τις αναλύσουμε στην συνεχεία. Ευχαριστώ. Κυρία Νίμπλερ. Thank you so much. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Είπατε ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σχετική νομοθεσία. Τι εννοείται γι' αυτό. για τις ρυθμίσεις των ε, συσκευών αυτών και των υλικών αυτών. Συμφωνώ. Δεν έχουμε λύση. Είμαστε στα χέρια των πολιτικών, της Κομισιόν και της βιομηχανίας για να βρει τους κανονισμούς. Μακροπρόθεσμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίζουμε μια ισχυρή νομοθεσία για το 3D printing, και όταν, δίδουμε, και όταν αντιμετωπίζουμε αυτούς τους εκτυπωτές όπως ένα οποιοδήποτε, μια οποιαδήποτε συσκευή, μέχρι να μεταβούμε πραγματικά στην ε, τρισδιάστατη ας πούμε, εκτύπωση, ε, τα μηχανήματα είναι ξεπερασμένα. Παραδείγματο χάρη, η λεπτή σκόνη, τα, τα λεπτά ορίματα, α πούμε, είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί πολύ. Θα πρέπει να βρούμε λύση. Για την ανακύκλωση δεν είμαι σίγουρο. Μέχρι στιγμή η συζήτηση είναι ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το 3D printing δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Γιατί χρησιμοποιούν πρόσθετα κτλ. Και τελικά το υλικό ε, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεν είναι απλό υλικό. Ε, έχει, για να γίνει το 3D printing, ας πούμε, έχει χρησιμοποιηθεί 100% ε, το υλικό. Στο μέλλον όμως, Το βασικό είναι να δίνουμε στα απόβλητα, να, πηγα... να καταλήγουμε στα απόβλητα πολύ απλά υλικά, ας πούμε. Πάντως σίγουρα ανακύκλωση δεν μπορεί να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο για να προσθέσει κάτι στη συζήτηση. Hello, good afternoon. Ε, Γεια σας. Να απαντήσω στις ανησυχίες σας πράγματι. Γίνονται εσωτερικές συζητήσεις ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες αυτές τις πτυχές. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ RDT, έρευνα ανάπτυξη, αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλε γενικέ διευθύνσει. Το πιο άμεσο σχόλιο μπορώ να κάνω είναι ότι αξιολογούμε αυτή τη στιγμή το διαγωνισμό, την προκήρυξη και υπάρχει ένα θέμα. Ε, ο στόχος είναι να ξεκινήσει ένα project που θα αντιμετωπίσει και τις τεχνολογικές αλλά, ε, προκλήσεις αλλά και τις μη τεχνολογικές πτυχές IPR, τυποποίηση, νομοθεσία, ρύθμιση κτλ. Και θέλουμε να λάβουμε υπόψη όσο, όλο το δυνα... ο, κατά το δυνατόν την ευρύτερη κοινότητα ε, ανοιχτής καινοτομίας και τρισδιάστατης εκτύπωσης. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσει την εργασία μας και θα έχουμε και πολλές ε, εκδηλώσεις, ε, εργαστήρια, σύντομα θα είναι όλοι οι εμπειρογνώμονες εκεί και, και εσείς είστε πρόσδεκτοι σε αυτή την εκδήλωση. Ε, Δεν μας λέτε και ποιος είστε. Είπατε είστε από τη έρευνα. Όνομα. Uh, my name is uh, Esteban. λέγομαι. Είμαι στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ RDT. Στην ε, ε ΔΕΛΤΑ τμήμα 2 για τις βιομηχανικέ τεχνολογίες. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε λάβει τη μελέτη, είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας, αλλά νομίζω διανεμήθηκε. Τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνετε στον ε, κύριο Ράινφελτ. Δεν θα σας απαντήσει. Ή όχι. Okay, will be answered. Θα σας απαντήσει. Μας το υποσχέθηκε. Δεν θα είναι εύκολο. Είμαστε σε καινούριο έδαφος εδώ σε ένα άλλο σύμπαν, βιομηχανική επανάσταση παρθυμών 5 εγώ θα έλεγα. Ε, και τέσσερα καλά θα ήταν να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσίαση και σε όλους και όλες εσάς ε, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τέλους μαζί μου εδώ. Και αύριο θα τα ξαναπούμε 9 το πρωί. Ευχαριστώ.